Bonjour chers collègues, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans la salle euh, de notre euh, commission. Nous allons commencer. Καλημέρα σας. Θα ξεκινήσουμε τις σημερινές μας πρωινές εργασίες με την κλασική διαδικασία, έγκριση δηλαδή της ημερήσιας διάταξης, διοτροποποίησης, ε, αναβολή της ακρόασης του κύριου Μπορκέντζιου και συνεδρία συντονιστών 2 και 4 απόγευμα. Σχόλια υπάρχουν για την ημερήσια διάταξη όχι και σας ευχαριστώ. Στο επόμενο θέμα. Le point suivant, που είναι η έγκριση των πρακτικών της 14ης Μαρτίου. Έχετε σχόλια, διορθώσεις, όχι και σας ευχαριστώ. Άρα εγκρίνεται, εγκρίνονται τα πρακτικά και ξεκινάμε την ακρόαση που έχουμε σήμερα το πρωί για την διασυνοριακή απόκτηση εκείνη της περιουσίας με τον καθηγητή Σπάρξ. 15 λεπτά σας παρακαλώ. Και σας καλώ ε, κατά τη διάρκεια της ομιλίας να ρίχνετε και μια ματιά στο ρολόι. Καλώς ήρθατε και με χαρά σας ακούμε. Καλημέρα σας, Πρόεδρε. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Το όνομά μου είναι Peter Sparks, καθηγητής στο δίκαιο το σχετικό με την ακίνητη περιουσία στο Southampton, ε, κάποτε λιμάνι από το οποίο ξεκινούσαν τα υπεροκειάνια προς την ε, Αμερική. Εκπρόσωπο. κονσόρτσιουμ που έχει σχηματιστεί από τον, κύριο, τον καθηγητή Ράναν από τη Βρέμη, τον Μαρτ και τον υποφαινόμενο, την Ταραγκώνα και την ε, Σιλισία της Πολωνίας. Έχουμε λοιπόν διερευνήσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ε, οι πολίτες όταν θέλουν να αγοράσουν ε, κατοικία σε κράτος μέλος άλλο από αυτό της ε, προέλευσής τους και κοιτούμε τα προβλήματα τα οποία τακτικά αντιμετωπίζει κανείς ως προς τις συναλλαγές σε περίπτωση που κανείς αγοράζει ένα εξοχικό σπίτι Φιλιππίνη στο εξωτερικό, αλλά και άλλα ασυνήθη προβλήματα. Κυρίως λοιπόν θα μιλήσουμε για, τη δεύτερη κατηγορία, αλλά αφού σας εκθέσουμε εν γέννη τα πρώτα, την πρώτη κατηγορία. Θέλω λοιπόν ιδιαίτερα να σας υπογραμμίσω εδώ τις λευκές γραμμές που βλέπετε στο χάρτη. Αυτές οι γραμμές στο χάρτη είναι τα εθνικά σύνορα των 28 κρατών μελών. Και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι δεν είναι μόνο 28 τα συστήματα έγκυας ιδιοκτησίας στην Ευρώπη. Φτάνουν τα 50 περίπου, γιατί η Ισπανία έχει χωριστεί νομοθεσία από την Καταλωνία, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο παρουσιάζει κοινό σύστημα για την ε, ε, Αγγλία και την Ουαλία με το Common Law, ενώ η ε, Σκοτία ακολουθεί το σύστημα του Ρωμαϊκού Δικαίου. Υπάρχουν ζητήματα επίσης αρμοδιοτήτων όπως προκύπτει από το άρθρο 347 της Συνθήκης για τη Λειτουργία. Έτσι λοιπόν έχουμε περιοριστεί μόνο στην εξέταση περιπτώσεων όπου είναι αδιαφυσβήτητε οι αρμοδιότητε, ε, σε περίπτωση δηλαδή υπερσυνοριακών συναλλαγών και αγορών περιουσιακών στοιχείων. Και θα παρακαλέσω τον δόκτωρα Ράλι να κάνει, να κάνει τη συνέχεια ε, την παρουσίαση των υπόλοιπων διαφανειών. Θέλουμε λοιπόν να κοιτάξουμε πόσοι είναι αυτοί καταρχάς οι οποίοι αγοράζουν ακίνητα στο εξωτερικό. Ε, δύσκολο έργο. Πολλοί είναι οι πολίτες που επιλέγουν να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα. Ε, κατηγορίες όπως εργαζόμενοι, όπως αυτοί που παραγωγούν μια δεύτερη κατοικία, συνταξιούχοι, αλλά και διαμεθοριακοί εργαζόμενοι, όπως συμβαίνει στην περιοχή γύρω από το Λουξεμβούργο, παραδείγματος. Μπορεί να είναι δύσκολο λοιπόν να υπολογίσουμε τα, ε, τον αριθμό των περιπτώσεων, αλλά θα έπρεπε τουλάχιστον τις συναλλαγές να μπορούμε να τις ε, διαγνώσουμε, αλλά και αυτό ήταν δύσκολο. Βεβαίω, ε, τα κτηματολόγια θα έπρεπε να είναι σε θέση να προσφέρουν τα στοιχεία αυτά για τι συναλλαγές έτσι ώστε και να, μην, ε, να καταγράφονται όλοι για να μην ε, διαφεύγουν του ελέγχου των εθνικών φορολογικών συστημάτων και πρέπει να βρεθούν συστημικές λύσεις για τα μεγάλα αυτά προβλήματα. Μια διαμεθοριακή λοιπόν αγορά ακινήτου. Βλέπετε εδώ δύο μεγάλα τετράγωνα ένα με χρώμα προς το μουσταρδί και ένα προς το πράσινο, δύο κράτη-μέλη δηλαδή. Στα δεξιά βλέπετε τη χώρα όπου, όπου βρίσκεται ο πολιτής του ακινήτου, αριστερά τη χώρα του αγοραστή. Το π σημαίνει αγοραστής, το β σημαίνει πολιτής και εμείς κοιτάμε την πτυχή περισσότερο του αγοραστή, από αυτό, αντίθετα από αυτό που συμβαίνει πολύ συχνά ε, όταν ο, ο νομικός δικηγόρος ή συμβολιογράφος εξετάζει την ε, αγοραπολισία, την κοιτάει συνήθως από την πλευρά του πολιτή. Εμείς λοιπόν κοιτάμε από την πλευρά του αγοραστή τα δεδομένα. Η σκούρα γραμμή με το βέλος, η οριζόντια γραμμή, μας δείχνει την φορά της συναλλαγής. Και η κατακόρυφη συμβολίζει τα σύνορα, την παραμεθόριο που διέρχεται κανείς κατά την αγοραπολισία. Και στο ανώτερο μέρος ε, της εικόνας βλέπετε ότι σχεδόν σε όλες τις χώρες απαιτείται η παρουσία δικηγόρου. Η ομάδα δείχνει το σύστημα το υπηρετικό ή του ρουμαϊκού δικαίου όπως λέγεται με παρουσία συμβολιογράφου του κράτους του πολιτή. Απαραίτητη. Φραγμή ή σύνορα. Εδώ έχετε Ωραία λοιπόν ως προς την διασυνοριακή αγοραπολισία ακινήτων. Ε, υπάρχουν πολλοί φραγμοί και όρια, πολιτική καταρχάς, πολιτικά όρια. Δεν υπάρχουν. Ένα Γερμανό μπορεί να αγοράσει στην Αυστρία χωρί ιδιαίτερε δυσκολίε. Η γλώσσα δεν αποτελεί πρόβλημα. Κατά κάποιον τρόπο ομοιάζει, λέει ο μιλητή. Και ο αγοραστή μπορεί να αντιληφθεί διαφορές που μπορεί να προκύπτουν στην συναλλαγή. Αλλά προβλήματα υπάρχουν. Αν ένας Βρετανός αγοράζει στην Ισπανία ένα ακίνητο. Πρώτα απ' όλα, γιατί υπάρχει διαφορά μεταξύ του ε, αγγλοσαξονικού και του ρωμαϊκού δικαίου, common law, civil law, οι διαφορές των ένωμων τάξεων δηλαδή. Μετά έχουμε την εμπλοκή συμβολεογράφου αντί για δικηγόρου, ως δεύτερη διαφορά. Και τρίτον, ε, μη οικία και αναπάντεχα ε, αναπάντεχη για τον αγοραστή διαδικασία. Η γλώσσα βεβαίως είναι ένα πρόβλημα, καθώς με ιδιαίτερη βέβαια έμφαση στην ειδική νομική ορολογία και ο συνάδελφος θα ασχοληθεί τώρα με τα θέματα των, ε, της ευρωπαϊκής αρμοδιότητας. Με αυτούς τους φραγμούς λοιπόν και προσπαθώντας να δώσουμε προστασία στο πλαίσιο αυτό οι περισσότερες ε, συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών έχουν να κάνουν συναλλαγές μεταξύ καταναλωτών όταν πρόκειται για αγορά κοινή του και όχι μεταξύ εμπόρου και ιδιώτη και καταναλωτή πιστεύουμε ότι πρέπει ε, παρά το γεγονό ότι μπορεί να έχουν καθαρά ιδιωτικό χαρακτήρα αυτέ οι συναλλαγέ, να εμπλέκεται και η ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά τι ασυνοριακέ πτυχέ τη ε, υπερμεθόρια αυτή ε, συναλλαγή. Υπάρχει κίνηση κεφαλαίων πέραν των συνόρων και θεωρούμε ότι εκείνο ο οποίο πάει σε μια άγνωστη χώρα να αγοράσει χρειάζεται υποστήριξη προκειμένου να στηριχθεί σε ένα ισότιμο πεδίο και επίση τα ζητήματα τη διαφήμιση, τη δράση των διαφημιστών ή των υπηρεσιών που προσφέρονται από τη νομική υποστήριξη, δηλαδή ε, η παροχή υπεσυνοριακη υπηρεσια έχουν μεγάλη σημασία. Ε, ιδιαίτερο ρόλο αναγνωρίζουμε σε σχέση με τα νεότευκτα ακίνητα, πολλά ε, εξοχικά, πολλές εξοχικές κατοικίες εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία και ιδιαίτερα εδώ έχουμε να κάνουμε συναλλαγές επιτοπλίστων εμπόρου προς καταναλωτή. Και εδώ ζητούμε λεπτομερή ενημέρωση, γλωσσικά δικαιώματα εξυπηρέτησης προς τη γλώσσα και βέβαια προσφορά νομικής υποστήριξης πριν οι αδίποτε βήματα σχετικά με τη συναλλαγή, κυρίως να πρόκειται για περίπλοκα και διαφορετικά νομικά συστήματα. Θα ξαναδώσω το λόγο τώρα στον Πίτερ για τις συστάσεις μας. Θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε σε σχέση με την αναρμόνιση των ε, δικαιωμάτων σε εκείνη την περιουσία, στην ε, ομοιόμορφη και πλήρη ενημέρωση του καταναλωτή σε σχέση με το τι αγοράζει. Έχουμε εντοπίσει δύο κατηγορίες πληροφοριών, δύο επίπεδα πληροφόρησης, ε, γενικές πληροφορίες και συγκεκριμένες ε, πληροφορίες ορόσημα και εδώ βλέπετε στις αγγίλες της συστάσεις μας στο τελευταίο, στο τελευταίο κεφάλαιο. Προτείνουμε το δικαίωμα στην, ενημέ, στην πληροφόρηση να προκύπτει ως δικαίωμα σε σχέση με γενικές πληροφορίες, τη διαφήμιση, του ακινήτου την τυποποιημένη ενημέρωση σε σχέση παραδείγματι με την οδηγία για, την, ε, για τις πιστοτικές συμβάσεις σχετικές με αγορά νεοτεύκτου κατοικίας και άλλες πληροφορίες σχετικές με την συναλλαγή, με τις συνθήκες συναλλαγής. Επίσης είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι γενικά Μπορεί να είναι ικανοποιημένοι οι καταναλωτές στην Ευρώπη από την υπηρεσία ε, που λαμβάνουν, καθώς ε, πολλά πράγματα πηγαίνουν πολύ καλά, αλλά υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν ε, προβλήματα, δεν καλύπτονται πάντοτε οι ανάγκες των καταναλωτών και γι' αυτό εμείς επιμένουμε να προσφέρονται οι βέλσες δυνατές πρακτικές και βεβαίως θα πρέπει να προσφέρουμε να προσφέρονται στο δυνατόν καλύτερη ενημέρωση σε σχέση με την ε, επιδίωξη πώληση πέραν των συνόρων. Θα πρέπει να συμπληρώνονται τα έντυπα κατά πλήρη τρόπο και όχι να αρκούμαστε σε μια ε, παρουσία στο γραφείο του συμβολογράφου εν ώψη της συναλλαγής. Η εκπρόσωποι των συμβολιογράφων λένε ότι δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα ή ότι θα χρειαζόταν μια τέτοια, μια τέτοια ε, παρέμβαση. Αλλά εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει πληρέστερη ενημέρωση και πολύ καλά κάνετε και έχετε την έκθεση αυτή και θα πρέπει να διερευνηθούν τα επίπεδα ικανοποίησης των καταναλωτών στις περσινοριακές ε, συναλλαγές που θα δείξουν πιστεύω πως παραμένουν τα προβλήματα. Βέβαια τα προβλήματα παραμένουν σε μια ε, μικρότερη σειρά περιπτώσεων, ωστόσο θεωρούμε πως όταν υπάρχουν έχουν να κάνουν με απουσία πλήρους υποστήριξης με νομικές συμβουλές. Ασφαλώς μπορεί να υπάρχουν συμβουλέ σε σχέση με την μεταβίβαση τη περιουσία, αλλά δεν είναι πάντα αρκετά λεπτομερής ω προς τις ε, λεπτομέρειε τη ε, σύμβαση ε, αγοραπολισίε ω προς το γενικότερο δίκαιο για την εγκατάσταση, τα οικογενειακά δικαιώματα, που είναι πολύ σημαντικά, ιδιαίτερα με τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ του αγγλοσαξονικού και του ρωμαϊκού συστήματος. Και νομίζω ότι τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ευρωβουλευτές είναι ότι δεν δίνονται πλήρες, πληροφορίε. πληροφορίες. Θα πρέπει πιστεύουμε να προσφέρεται ευρύτερη ενημέρωση στον τομέα αυτών και για να κλείσω υπάρχουν κάποιες ε, ακραίες περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν και όπου Φαντάζομαι πως ε, οι αγοραστές απέφθηναν ε, τα αιτήματά τους σε ευρωβουλευτές ε, για κάποιες ασυνήθιστες καταστάσεις που καταγράφονται εδώ στη διαφάνεια. Θα τα γνωρίζουν οι ευρωβουλευτές σας. Και κάποιες τελικές παρατηρήσεις. Ο δικηγόρος δεν μπορεί να προφλέξει κανέναν κατά της αλλαγής της νομοθεσίας. Όταν κατά τη στιγμή της αγοραπολισίας υπάρχουν προβλήματα, πρέπει η νομική συμβουλή και έρευνα από το δικηγόρο να εξασφαλίζει ότι δεν ε, έχει ελαττώματα αυτή η συναλλαγή, αυτή η σύμβαση. Πρέπει η δυνάμη του 345 που επικαλέστηκα και νωρίτερα να ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα προβλήματα αυτά. Κάποια από τα προβλήματα έχουν να ε, κάνουν κατά πάσα πιθανότητα και με την παρεμπόδιση του βασικού δικαιώματος για μεταφορά κεφαλαίων, ιδιαίτερα στην περίπτωση των μη φανερών υποθηκών στην Κύπρο, όπου δεν έχει ο ε, αγοραστής πλήρη απόκτηση τίτλου για τα χρήματα που έχει πληρώσει. Επίσης, στην περίπτωση της Βαλένσια είχαμε ζητήματα με απαλωτρίωση γεών και μας ξαφνιάζει το γεγονό ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν έχει προσφέρει επαρκείς λύσεις στο πρόβλημα αυτό. Ελάχιστες ε, είναι μάλιστα οι δίκες που έχουν ε, ξεκινήσει από Ισπανούς ή από την Ισπανία ως χώρα προς το δικαστήριο του Στρασβούργου για να αμφισβητήσουν αυτές τις απαλωτριώσεις. Υπάρχουν λοιπόν ε, ζητήματα που μπορούν να προαχθούν, ε, υπάρχουν εκκρεμότητες, είναι δύσκολο να δοθούν οι λύσεις στο πρόβλημα. Πολλές όπως περιπτώσεις πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί με σωστές συμβουλές από το δικηγόρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά δεν έχει την αρμοδιότητα για την εναρμόνιση των συστημάτων ε, έγκυας ιδιοκτησίας και θα πρέπει να εξετάσει τι μπορεί να κάνει για να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci Σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, εξηγήσεις αυτές ο Τιερι Βασχό, υπεύθυνο τη Οργάνωση Συμφωλιογράφων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, θα πάρει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωκοινοβούλιο και την Επιτροπή σας που μας δίνει την δυνατότητα να σχολιάσουμε τη μελέτη αυτή. Οι Ευρωπαίοι Συμβολιογράφοι σημειώνουμε τα απορίσματα της μελέτης και βέβαια δεν έχουμε επί της αρχής καμία ε, διαφωνία σε ό,τι αφορά την ε, μελέτη αυτή που ανατέθηκε από ε, το Κοινοβούλιο σε αντίθεση από αυτά που ο καθηγητής Σπάρξ στην αρχή. Πάντως θα ήθελα να κάνω κάποιες αρχές παρατηρήσεις και επιφυλάξω ό,τι αφορά το περιεχόμενο. Η νομική προσέγγιση είναι κάπως ε, κατά προσέγγιση και κάποιες φορές περιέχει σφάλματα. Οι συμβολογράφοι θεωρούμε ότι τα σφάλματα αυτά θα μπορούσαν ενδεχομένως να είχαν αποφευχθεί αν εν λόγω μελέτη συνοδευόταν, μάλλον είχε ε, γίνει από ένα πάνελ ειδικών που θα εκπροσωπούσαν περισσότερο και γεωγραφικά ε, την Ευρώπη και σε ό,τι αφορά του επαγγελματίες του κλάδου. Δεν την περίμετρο αυτή τη μελέτη, πολύ συχνά θεωρούμε ότι περιστρέφεται γύρω από ζητήματα απόκτηση από Βρετανού έπικο προ την Ισπανία. Ε, ακούσαμε πρόσφατα το παράδειγμα αυτό και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα ε, όμως τα οποία θα έπρεπε να είχαν υπογραμμιστεί και τα οποία θα αφορούσαν και χώρες ε, ε, πιο συγγενείς σε ό,τι αφορά το δίκαιο, παραδείγματος χάρη Γαλλία, Ισπανία. Επίσης, σε ό,τι αφορά την επιστημονική και νομική βιβλιογραφία, πολλές φορές γίνονται αναφορές. Επίσης, σε κάποιες εκφράσεις που λένε wishing, δηλαδή δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρα και κατηγορηματικά αυτά που αναφέρονται. Επίσης θεωρούμε ότι υπάρχουν νομικές μελέτες, στατιστικές, βάση, τεκμηρίωσης, βιβλιογραφία σημαντική. Θα έπρεπε και εμείς να είχαμε δώσει τις ε, απόψεις μας. Ο κύριος Σπάρξ, ο καθηγητής και η ομάδα του θα είχαν πιστεύω επωφεληθεί. Επίσης ε, λυπούμαστε που ε, το επάγγελμά μας αντιμετωπίζεται βιβλιογραφικά με κάποιες επίσης εκφράσεις όπως comic, nightmare, hot, κάπως υποτιμητικά θα έλεγα μας αναφέρουν. Ε, πρέπει να σας πω όμως ότι εμείς ε, ε, είμαστε στο πλευρό των Ευρωπαίων πολιτών 100% σε ό,τι αφορά αυτές τις συναλλαγές, τις συνεργές απόκτησα κινήτων. Έχουμε πρόβει σε κάποιες διαπιστώσεις, έχουμε κάνει προτάσεις για βελτιώσεις όπου Συμβούλιο, Κοινοβούλιο, υπηρεσίες τους θα μπορούσαν να βελτιώσουν ίσως κάποιες από αυτές τις συναλλαγές. Υπάρχει ενημέρωση συνεχής και στην ιστοσελίδα μας δίνουμε πληροφορίες εδώ και κάποιους μήνες για όσους θέλουν να αγοράσουν ένα κίνητο ε, στις 22 χώρες μέλη που έχουν ε, τις υπηρεσίες αυτές. Έχουμε και την πλατφόρμα ε, συνεργασία συμβολογράφων Φίντες που μπορούν οι πολίτες να συμβουλευτούν μέσα αυτής της θέση του πολλούς επαγγελματίες όταν πρόκειται για τις ε, συναλλαγές κινήτων, ακινήτων, ε, αγοραπολίσεις ακινήτων και βέβαια σε πολλές χώρες μέλη διατίθεται δωρεάν πληροφορίες πολίτες ε, για το νομικό σύστημα της χώρας και πραγματικά καταβάλλονται και προσπάθειες ε, σημαντικές για να μεταφραστούν τα σχετικά έγγραφα στα αγγλικά. Αυτό το οποίο θέλουμε να επαναλάβουμε είναι ότι προσφέρω, είμαστε στη διάθεση ε, για συνεργασία. Νομίζουμε ότι υπάρχουν ε, περιθώρια βελτίωσης. Ε, το είπε και ο καθηγητή Σπάρξ βέβαια ότι οι συναλλαγές αυτές γίνονται ομαλά, δεν θα πρέπει απλά να εστιάσουμε σε λίγα προβλήματα. Μπορεί να είναι λυπηρό το ότι υπάρχουν, αλλά νομίζω Στι περισσότερε περιπτώσει αυτά τα προβλήματα ανήκουν στο παρελθόν. Είμαστε στη διάθεση λοιπόν, όπω είπα, του Κοινοβουλίου, των Ευρωπαίων πολιτών για να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε ε, το σύστημα διασυνοριακών αγοραπολισιών ακινήτων. Ευχαριστώ, Πρόεδρο. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και του ε, ε, προηγούμενου ομιλητέ. Οι συνάδελφοί μα έχουν ερωτήσει. Παρακαλώ, εσεί. Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν έχω ερωτήσει. Θα ήθελα η μελέτη να είναι πιο ενδελεχή. Θα κάνω κάποιε παρατηρήσει. Ακούσαμε ότι δεν υπήρξε διαβούλευση ή επαφή ανάμεσα στους προσώπους των συμβολιογράφων και σε αυτούς που ανέλαβαν τη μελέτη. Είναι πολύ δύσκολο να εμπιστευτούμε μία μελέτη που έγινε σε ένα γραφείο, σε απομόνωση, χωρίς καμία επαφή με τους άμεσα εμπλεκόμενου στο θέμα αυτό, ε, ούτως ώστε να λάβουν χώρα αυτές οι διασυναριακές αγορές. Σε ό,τι αφορά τα λεγόμενα φράγματα, πέρα από τα γλωσσικά ή φράγματα ή προβλήματα, οι διαδικασίε είναι διαφορετικέ. Και μάλιστα θα μπορούσαμε να δούμε τις διαδικασίες ως δίκτυα ασφαλείας που χρειάζεται ο αγοραστής όταν αγοράζει ακίνητο σε ένα διαφορετικό κράτος μέλος. Αυτό το δίκτυο ασφαλείας εξασφαλίζεται από τον δικηγόρο στο Ηνωμένο Βασίλειο ή από το συμβολιογράφο σε άλλα κράτη-μέλη που αναλαμβάνει όλε τι απαραίτητε διαδικασίε, ούτω ώστε να ξέρει ότι είναι ασφαλή ο αγοραστής. Εγώ ήρθα σε επαφή με τι βελγικέ αρχέ Για να αγοράσεις ε, ένα κίνητο στο Βέλγιο χρειάζεστε μια περιοδο δυο δύο-τριών μηνών μέσα στην οποία ο συμβολιογράφος ελέγχει διάφορα πράγματα ούτω ώστε να εξασφαλίσει ότι με την αγορά αυτού του ακινήτου δεν θα έχει κανένα πρόβλημα και ότι είσαι ο πραγματικό αγοραστή. Καλό θα ήταν λοιπόν η μελέτη αυτή να έχει γίνει με τη συνεργασία των συμβολιογράφων, γιατί αυτοί εξασφαλίζουν αυτές τις αγορές. Κυρία Ρέινερ και συνεχεία ο κύριος Μάντες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, εκ μέρους ε, ε της Ευρωπαϊκής ε, υπηρεσίας των ειδικών ε, του κλάδου. Θα θέλαμε να σχολιάσουμε και εμείς. Θα θέλαμε και εμείς να κάνουμε τα σχόλιά μας. Σε ό,τι αφορά αυτή τη μελέτη λοιπόν ε, για τις διασυνοριακές οραπολισίες ε, ακινήτων, ιδίως σε ό,τι αφορά ακριβώς αυτό το πλάτο της ακίνητης περιουσίας, την αποκτήση ακινήτων, αναφέρονται κυρίως περιπτώσεις αγροπολισιών ακινήτων μεταξύ ε, Ηνωμένου Βασιλείου και Ισπανίας. 14% ε, του συνόλου ε, των συναλλαγών αυτών γίνονται από ξένους υπηκόους και το 16% από Βρετανούς. Κάποιες παρατηρήσεις απλά. Φυσικά και είμαστε στη διάθεσή σας για να αναλύσουμε αυτή τη μελέτη. Πρώτες μας σκέψεις πάντως είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο θα έπρεπε να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό. Υπάρχουν συμφωνίε μεταξύ κρατών μελών και νομίζω ότι τα προβλήματα επιλύονται με αρκετά ευέλικτο τρόπο και δεν είμαστε βέβαιοι κατά πόσον ε, θα έπρεπε να ε, βρούμε λύσεις που τελικά θα κάνουν πιο δίσκαμπτες και θα δυσχεράνουν περισσότερο αυτές ε, τις ροές, αυτές τις συναλλαγές. Επίσης, σε ό,τι αφορά κάποιες ανακρίβειες ε, για κάποια συστήματα, το ισπανικό σύστημα είναι δημόσιο και βασιζόμαστε στην ε, ε, καταγραφή και στη δήλωση των, και όχι στην αντιπαραβόλη όπως είναι το γαλλικό σύστημα. Επίσης θεωρούμε ότι αυτό που λέγεται ότι τα προβλήματα και τα όρια θα πρέπει να δίνονται πληροφορίες στα κτηματολόγια και να μελετούν τα κτηματολόγια. δεν υπάρχουν σε όλε τι χώρε πρώτον κτηματολόγια και δεν δίνουν τα κτηματολόγια όλες αυτές τις πληροφορίες. Στις περισσότερες συναλλαγές δεν προκύπτουν κάποια προβλήματα, σε κάποιες μπορεί. Επίσης, γίνεται αναφορά σε κάποια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι ε, αγοραστές. Όμως ε, τα προβλήματα αυτά τα αντιμετωπίζουν όλοι οι αγοραστές ε, της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Το πρόβλημα προκύπτει από το βαθμό στον οποίο σε ό,τι αφορά τους αγοραστές θα πρέπει να περτερούν κάποια ε, δικαιώματα του κράτους ε, και να επηρεάζουν κάποιες εθνικές πολιτικές. Και ποια είναι τα... Ποιες είναι οι πληροφορίες οι οποίες μπορούν να δίνονται στους πολίτες. Αυτό επαναλαμβάνω όμως δεν είναι ζήτημα που αφορά μόνο τους αλλοδαπούς αγοραστές αλλά και τους ε, ντόπιου. Σε ό,τι αφορά τώρα ένα πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με το ότι δεν είναι γνωστά, δεν είναι γνωστοί οι κανόνες δημόσιου δικαίου θα μπορούσαν να επηρεάσουν ε, τις διάφορες συναλλαγές, θεωρούμε ότι πέραν των προβλημάτων ε, που μπορεί να προκύπτουν τα διάφορα τόκια της καταγραφής, Υπάρχουν ζητήματα με την αρχαιοδότηση και την καταγραφή στην Ισπανία πρόκειψαν κάποια προβλήματα, αλλά έχουν ε, γίνει απαραίτητε τροποποίησεις. Σε ό,τι αφορά τώρα τις προτάσεις για τους ε, αλλοδαπούς αγοραστές, αναφέρονται κάποια, κάποιες αμφιβολίες σε σχέση και με την εμπειρία των ξένων αγοραστών στην Ισπανία αλλά και μας εκπλήσει το γεγονός ότι υπάρχει το Ήμολα, ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει και έργο πίσω του, είναι ένα έργο διασύνδεσης των Ευρωπαϊκών Υποθυκοφυλακίων, αλλά δεν γίνεται σε αυτό καμία, σε αυτή την μελέτη, καμία μία σε αυτό το αρχείο. Σίγουρα υπάρχουν ε, κάποια όρια στην παρέμβαση Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για διασυνοριακές συναλλαγές και ίσως εκεί θα μπορούσαμε να... Ε, Φαντάζομαι θα μπορούσαν να ε, υπάρχουν κάποιοι κανόνες σε επίπεδο ευρωπαϊκό για την προστασία των καταναλωτών, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς. αν αυτό που λέγεται στην έκθεση φωτοκόμες κλώσ, αν αυτό που υπάρχει στον Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να υπάρχει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τα μελετήσουμε και θα σας δώσουμε γραπτό στα σχόλιά μας, αλλά βέβαια σίγουρα είμαστε στη διάθεσή σας για να ε, συνεργαστούμε και σας ευχαριστούμε πολύ εμείς οι υποθηκοφύλακες. Merci à vous. La parole est à Madame Regner. Ευχαριστώ κυρία Ρέγνερ, και μετά η κυρία Στέλλα Σφυραγκούτ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ για την παρουσίαση της μελέτης. Είναι πολύ ε, διεξοδική. Πρέπει να τη διαβάσουμε μεγάλη προσοχή για άλλη μια φορά. Πάντως μέχρι τώρα ευχαριστώ για την παρουσίαση και θέλω να κάνω τις εξή παρατηρήσεις. Καταρχάς είναι πολύ σημαντική αυτή η δουλειά. Ως προς την πρόσβαση πάντως θέλω να επισημάνω τα εξή συμπληρωματικά. Ε, η διαμονή είναι η κατοικία καλύτερα είναι βασική ανάγκη και όχι υπηρεσία. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να τη δούμε και υπό το φως των τεσσάρων ελευθεριών, βέβαια και της ελευθερής κυκλοφορίας των κεφαλιών στην Ευρώπη, αλλά επαναλαμβάνω ότι πρόκειται για θεμελιώδη ανάγκη. και σε πολλές χώρες αναγνωρίζεται το δικαίωμα στην κατοικία και ως οικουμενική υπηρεσία που πρέπει να εγγυάται το κράτος. Και βέβαια σε αυτό υπάρχει και η ευθύνη να μην επιτραπεί υπερβολική άνοδος των τιμών. Σε αυτό, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη σε κάθε αντίστοιχη μελέτη και τα συμπράσματα που απορρέουν από αυτήν. Υπάρχουν ε, ε, κράτη επίσης τα οποία οι πάντες είναι ιδιοκτήτες, πάντοτε αγοράζεται δηλαδή η ιδιοκτησία, ενώ άλλα κράτη στα οποία επιτοπλίστων ε, μένει κανείς σε μισθωμένη κατοικία. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, αντιπαραθέσεις παραδείγματι μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάτω χωρών ως προς τα οικονομικά επίπεδα και όρια, ανώτατα όρια του, της κοινωνικής στέγης ή της στέγης που μπορεί να είναι ανεκτή ε, κοινωνικά. Επίσης, θέλω να ρωτήσω τα εξή, Εάν υπάρχουν από πλευράς των κρατών μελών, ε, αν υπάρχει δεδηλωμένο ενδιαφέρον για την παρακολούθηση αυτών των κινήσεων των ακινήτων και θέλω να δω από τη μελέτη σας αν έχετε κάτι και επίση από τα συστήματα των οικοφυλακίων ή καλύτερα των κτηματολογίων που είναι πολύ διαφορετικά στην ε, Ευρώπη. Στην ε, Αυστρία βεβαίως έχουμε ένα σύστημα κτηματολογίου με πολύ διαφορετικά όμως στοιχεία και το ξέρουμε πολύ καλά, το είδα μάλιστα και με την κρίση στην Ελλάδα τη σχετική, ότι είναι πολύ διαφορετικά τα συστήματα και οι εγγραφέ, δηλαδή ποια δικαιώματα εγγράφονται, πώς περιγράφονται μέσα στο κτηματολόγιο κτλ. Και πώς αναγνωρίζεται βέβαια το ε, τεμάχιο γης. Θα ήταν καλό λοιπόν σε μια τέτοια μελέτη και το ανέφερε και ο συνάδελφος από το ΕΛΚ ε, να ε, προβάλλεται ιδιαίτερο η ανάγκη για την ασφάλεια δικαίου για τον αγοραστή ενός ακινήτου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και ιδιαίτερα πρέπει να το προστατεύσουν οι συμβολεογράφοι, εκείνοι οι οποίοι έχουν το κύριο έργο στην παροχή των σχετικών συμβουλών. Οι συμβολεογράφοι λοιπόν έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Εστέρα Σφαρακούτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, καταρχάς. Ήταν μια καλή πρωτοβουλία το να φτιάξουμε μια έκθεση για το τι αντιμετωπίζει ένας Ευρωπαίος πολίτης όταν αγοράζει ακίνητα σε άλλο κράτος μέλος και να δούμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας βέβαια και να δούμε πού ακριβώς υπάρχουν τα προβλήματα, πού έγκυται τα προβλήματα. Συμφωνώ με το συνάδελφο από το ΕΛΚ και το συνάδελφο από τους σοσιαλιστές θα πρέπει όταν κάνουμε μια τέτοια μελέτη, στην πραγματικότητα να ερχόμαστε σε, να επαφή και με τους συμβολιογράφους και με τους υποθηκοφύλακες, γιατί αυτοί είναι οι επαγγελματίες οι οποίοι εξασφαλίζουν τις διασυνοριακές συναλλαγές και αγορές. Και αυτοί μας δίνουν τη βεβαιότητα ότι όλα γίνονται με βάση το πνεύμα και το γράμμα του νόμου. Ο εκπρόσωπος των υποθηκοφυλάκων είπαν ότι υπάρχουν μία σειρά από θέματα ε, προβληματικά, ειδικά για την περίπτωση της Ισπανίας που αναφέρατε στην, έκθεση, στην μελέτη αυτή και επομένως είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη σας τι είπαν οι συμβολιογράφοι όσο και οι υποθηκοφύλακες. Κυρίως αναφέρεται σε ένα νόμο της Βαλένθιας ε, που πέρασε πριν από 10 χρόνια Το 2014 όμως έγινε ένας νέος αστικός νόμος ε, όπου τον στήριξαν οι περισσότερες ε, πολιτικές δυνάμεις. Είχαμε πολλά προβλήματα στις ακτές της ε, Βαλένθιας και η Επιτροπή Αναφορών ζήτησε, έλαβε πάρα πολλά παράπονα και ζητήθηκε να γίνει μία τροποποίηση του νόμου για να προστατευτεί και το περιβάλλον και η ιδιωτική περιουσία. Ε, και το 2014 έγινε μια τροποποίηση του νόμου αυτού, του παλιού νόμου. Στην περίπτωση μπάση πτώση της Ισπανίας πρέπει να σας πούμε ότι πρόκειται ε, για ένα δημόσιο σύστημα. Υπάρχει αυτό το σύστημα των υποθηκοφυλακίων στην Ισπανία. Ε, υπάρχει ένα συντονισμό ανάμεσα στου ε, συμβολιογράφου, δηλαδή ο συμβολιογράφο έρχεται σε επαφή με τον υποθηκοφύλακα για να ανοιχτευτούν πιθανά προβλήματα στην αγορά του ακινήτου. Σα ευχαριστώ για τι ε, για τις ιδέες σας, τις ε, σας. Δεν, δεν ζητάει κανένα άλλο το λόγο. Θα περάσουμε στο επόμενο σημείο που αφορά τους ευπαθείς ενήλικες στην Ευρώπη. Θα δώσουμε το λόγο πάραυτα σε δύο άτομα και συνεχεία στη συναδελφό μας. Ο κύριος Γιάν Κάρισον. Έχουμε συνολικά ένα τέταρτο για αυτό το θέμα. Εν συνεχεία πρέπει να περάσουμε στην επόμενη ακρόαση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω τα πορίσματα της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δυνατότητα ε, των νομικών εργαλείων που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατεύσει τους ευπαθείς ανήλικες, ενήλικες συγγνώμη, στην ε, Ευρώπη. Ο παγκόσμιος ε, έχει ράσκει και ζει περισσότερο χρόνο. Έχουν γίνει εκτιμήσεις ότι μέχρι το 2025, 50, άτομα άνω των 65 ετών θα είναι το 35% του πληθυσμού με πάνω από 10% του πληθυσμού να είναι πάνω από 80. Καθώς το προσδόκιμο ζωής θα αυξάνει όλο και περισσότερο, θα αυξάνονται και οι αρρώστιες, όπως το Αλτσχάιμερ και η άνοια. Επίσης, ο παγκόσμιος πληθυσμός από την άλλη γίνεται όλο και πιο κινητός όλο και ταξιδεύει περισσότερο. Ο αριθμός στην Ευρώπη των ανθρώπων που ταξιδεύουν από χώρα σε χώρα αυξάνεται. Αυτές οι δύο τάσεις μαζί ε, αύξησαν τα διασυνοριακά προβλήματα που συνδέονται ε, με τη μετακίνηση και την ε, μεγάλη ηλικία. Κάνουμε αυτή τη μελέτη για να μελετήσουμε το αν θα ήταν δυνατόν και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει προστιθέμενη αξία ε, στην προσπάθεια επίλυσης αυτών των προβλημάτων. Η έκθεση που συντάχθηκε είναι η βάση για αυτή την παρουσίαση. Η έκθεση έχει πέντε κεφάλαια και η βασική εστίαση ε, αφορά τις εξηγήσει για τις ελλείψεις του τρέχοντος πλαισίου μαζί με την προστασία που δίδεται ε, από την ε, Σύμβαση Προστασίας της Χάγης του 2000. Καταρχάς, ας μιλήσουμε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Τι είναι αυτό το θέμα που μας απασχολεί. Για να δούμε τις κοινωνικές επιπτώσεις. Να πούμε το εξή παράδειγμα. Φανταστείτε ότι έχετε έναν Ιρλανδό που ζει στην Ελλάδα. Έχει περιουσιακά στοιχεία στην Ιρλανδία, αλλά μένει σε ένα διαφορετικό κράτος μέλος και γυράσκει και θέλει να επιτρέψει στον γιο του να διαχειριστεί την περιουσία του στην Ιρλανδία. Ε, δίνει λοιπόν, κάνει ένα πλεξούσιο στην Ελλάδα, ούτω ώστε να δώσει στο γιο του αυτή τη δυνατότητα να το κάνει. Αυτό το πλεξούσιο που συντάχθηκε στην Ελλάδα ισχύει στην Ιρλανδία. Ένα άλλο παράδειγμα ε, μπορεί να φωτίσει αυτό το πρόβλημα. Φανταστείτε ότι έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι Ούγγρος και που πεθαίνει στην Ισπανία. Ε, έχει την κόρη του, η οποία ζει στη Γαλλία, αλλά έχει ψυχολογικό ψυχικό πρόβλημα και βρίσκεται σε ειδικό ίδρυμα με βάση τα όσα επέβαλαν οι γαλλικές αρχές. Η γαλλική απόφαση ισχύει στην Ισπανία. Γιατί? Το θέμα είναι, μπορεί αυτή να αποδεχτεί την κληρονομιά που βρίσκεται στην Ισπανία. Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα, σε τέτοιου τύπου προβλήματα, εξαρτώνται από τις νομικές υποχρεώσεις που έχουν τα διάφορα κράτη-μέλη που εμπλέκονται. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν το τρέχον πλαίσιο που ισχύει εδώ. Πρέπει να δούμε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ κατακαιρματισμένο. Έχουμε διάφορα, διάφορους φορείς που εμπλέκονται. Στην αρχή είδαμε τη σύμβαση της Χάγης, την ε, ε, διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο και τη Σύμβαση Προστασίας των Ενηλίκων του 2000. Ε, υπάρχουν και πάρα πολλά όμως νομικά κείμενα που επηρεάζουν. Έχουμε την Σύμβαση που αφορούν τα μέτρα προστασίας από τη διάσκεψη της Χάγης. Έχουμε την Σύμβαση της Χάγης του 1978 και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία του 2006 που υπάρχει επίσης στην ατζέντα για τη σημερινή συνεδρίαση. Επίσης έχουμε και διάφορα άλλα μέσα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ε, το κανονισμό των Βρυξελών, τον κανονισμό της Ρώμης, έχουμε τον κανονισμό για τις κληρονομιές, τον κανονισμό για την προστασία και διάφορα άλλα εργαλεία. Όμως, κανένα από αυτά τα εργαλεία δεν ασχολείται συγκεκριμένα με το πρόβλημα της προστασίας των ευπαθών ενηλίκων και τα περισσότερα ευρωπαϊκά εργαλεία αποκλείουν τα θέματα της ικανότητας, ε, και αποκλείουν δηλαδή τους ανθρώπους αυτούς από τη συζήτηση και την προστασία. Υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν τα αποδεικτικά στοιχεία και που επηρεάζουν οριακά απλώς το θέμα μας. Επομένως, έχουμε μια πλειάδα από εργαλεία, έχουμε κατακαιρματισμό ε, διάφορους που εμπλέκονται σε αυτό το τομέα και λόγω αυτού του κατακαιρματισμού ε, και των διαφορών έχουμε διάφορα προβλήματα ε, αλληλεπιδράσεων ανάμεσα σε αυτά τα νομικά κείμενα. Και τα εργαλεία που υπάρχουν σε διεθνέ επίπεδο έχουν ε, πλήττονται από πολύ λίγες επικυρώσεις. Ο οργανισμός της Χάγης έχει επικυρωθεί από τρεις ευρωπαϊκές χώρες και την Αργεντινή. Επομένως, ενώ έχουμε κάποια εργαλεία που θα μπορούσαν να επηρεάσουν, στην πραγματικότητα έχουν πολύ περιορισμένη επίπτωση. Μόνο ένα συγκεκριμένο εργαλείο που ασχολείται με αυτά τα θέματα, η Σύμβαση Προστασίας των Ενηλίκων της Χάγης του 2000, είναι βασικά ε, το βασικό μας εργαλείο. Και αυτό αναλύουμε στην ε, κειμένη. Στις 13 Ιανουαρίου του 2000 υιοθετήσαμε τη Σύμβαση και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2009. Μόνο εννέα χώρε έχουν επικυρώσει αυτή τη σύμβαση αυτή τη στιγμή. Η Αυστρία, η Τσεχία, η Εστονία, Φιλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία και Σκοτία εντό του Βασιλείου και από τι 4 Μαρτίου του 2016 και το Μονακό. Άλλα αυτά κράτη-μέλη έχουν υπογράψει τη σύμβαση, αλλά δεν την έχουν επικυρώσει. Η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, Λουξεμβούργο και Ολλανδία και η Πολωνία. Η έκθεση ασχολείται με τους έξι αυτούς τομείς και ο πρώτος τομέας αφορά τους ορισμούς που έχει η σύμβαση. Το δεύτερο τμήμα μιλάει με τα διάφορα κομμάτια της σύμβασης, ε, του διαφόρου των τομέων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και το θέμα της συνεργασίας. Ένα βασικό θέμα είναι τα υποχρεωτικά πιστοποιητικά ή το θέμα του πληρεξούσου δικηγόρου και τα ελλείμματα που υπάρχουν εκεί. Να σας επιστήσω την προσοχή σε διάφορα προβλήματα που εντοπίστηκαν με βάση την έκθεση. Ένα από τα θέματα που αναφέρει ο ορισμός είναι ο ορισμός ε, μιας ε, βλάβη, ζημία που έχει κάποιο, ε, προβλήματο ψυχικού ή πνευματικού ή ανικανότητα. Ανικανότητα λοιπόν για δικαιοπρασία. Αν κάποιο, α πούμε, ε, είναι θύμα ε, τροχαίου στην Αυστρία, και δεν μπορεί να περπατήσει, ε, είναι σε ένα πυρικό καροτσάκι. Ο αδερφός της έχει ένα πλειοεξούσιο το θέμα είναι, αυτό το πληρεξούσιο ε, καλύπτεται από αυτή τη σύμβαση. Ήρθαμε σε επαφή με κάποιου συμβολιογράφου και με κάποιου ε, ειδικού και επαγγελματίε. Υπάρχουν προβλήματα με αυτόν τον ορισμό. Γιατί το ίδιο το άτομο δεν είναι κατά ανάγκη ευπαθέ, αλλά μπορεί να έχει ένα πρόβλημα πούμε, ε, και δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε νομική προστασία σε ένα άλλο κρατό μέλο. Αντίστοιχα προβλήματα έχουμε στο πληρεξούσιο όταν το άτομο το ίδιο δεν έχει πρόβλημα, αλλά το πρόβλημα προκύπτει αργότερα. Δηλαδή, τη στιγμή που συντάσσεται το πλειοεξούσιο, δεν υπάρχει πρόβλημα στο άτομο, αλλά αργότερα αποκτά. Επίσης, άλλα προβλήματα μπορεί να ανακύψουν. Και τα κατηγοριοποιούμε σε δύο βασικές κατηγορίες προσωρινά προβλήματα που επιλύονται αν όλα τα κράτη-μέλη ε, επικυρώσουν αυτή τη σύμβαση για προστασία των ενηλίκων και τα προβλήματα που θα παραμείνουν ε, ακόμα και αν όλα τα κράτη-μέλη επικυρώσουν τη σύμβαση. Τα θέματα που θα εξακολουθήσουν να παραμείνουν ακόμα και να επικυρωθούν από όλα τα κράτη-μέλη λοιπόν ε, υπάρχουν πολλά τέτοια προβλήματα το είδος της ε, ευπάθειας, τα ίδια τα μέτρα, ε, η αναγνώριση και το θέμα του πιστοποιητικού. Η ευρωπαϊκή δράση είναι πιθανή βάσει του νομοθετικού πλαισίου. Έχω ένα λεπτό βλέπω. Και το θέμα της επικουρικότητας επίσης αναφέρεται στην έκθεση. Ε, η νομοθετική βάση αναφέρεται με βάση το άρθρο 81, 2α, B, C και F. Και ο κανονισμός είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε, για να συμπληρώσουμε την επικύρωση της, ε, της σύμβασης της Χάγης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρον και ζητώ. Συγγνώμη που σας πίεσα, η κυρία Ζωελόν πρώτα και μετά η κυρία Μπερζογόν. Πέντε λεπτά εκάστε παρακαλώ. Όχι, ο συνάδελφός σας. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστώ την Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων γιατί μας επιτρέπει στην κυρία Λόν και εμένα να κάνουμε την παρουσίαση της μελέτης μας με τα κύρια ευρήματά της. Εντοπίζουμε, δύο κύρια αισθήματα, δηλαδή εάν το νομικό πλαίσιο που ισχύει αυτή τη στιγμή για την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρκεί και αν όχι τι, και αν ναι, τι είδους μέτρα, τι περιεχόμενο μπορεί να έχουν τα μέτρα που προβλέπονται κοιτάμε πρώτα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διεθνή προστασία των ε, ενηλίκων ε, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερος αξιολόγηση πλέον εκτιμάτων και δυναμικού της ε, Σύμβασης της ΧΑΙΚΣ του 2000 για τη Διεθνή Προστασία Ενηλίκων με βάση ανάλυση πρακτικών περιστατικών, ε, θεωρητική ανάλυση και ε, συνεντεύξεις με τους νομικούς που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Στη Γαλλία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο κοιτάξαμε την κατάσταση. Ιδιαίτερος φαίνεται να είναι αντιπροσωπευτική η κατάσταση στις αυτές χώρες για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Γαλλία έχουμε την κύρωση ήδη της ε, Χάγης μαζί με την Εστονία, την Φινλανδία, την Τσεχία και την Αυστρία. Η Ιταλία δεν δεσμεύεται από τη συνθήκη, από τη σύμβαση και εφαρμόζει το εσωτερικό δίκαιο, ιδιωτικό και διεθνές. Όπως άλλωστε, και η όπως άλλωστε και η Ιταλία και άλλες χώρες δεν έχουν κυρώσει, όπως το Βέλγιο, κατοχώρες, Πολωνία, Ισπανία. Το Ηνωμένο Βασίλειο από πλευρά του έχει ιδιαιτερότητες καταρχάς λόγω της νομικής του παράδοσης διαφορετικής από αυτή της Ιταλίας και της ε, Γαλλίας και ε, δεύτερον διότι έχει μια μεικτή προσέγγιση εναντί της Σύμβασης της Χάγης έχει κυρώσει μεν τη Σύμβαση η Σκοτία ενώ η, Αγγλία, η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία προτιμούν να μην ε, γίνουν συμβαλόμενα μέρη στη Σύμβαση της Χάγης. Βλέπουμε λοιπόν ε, πρακτικές δυσκολίες σε σχέση με την διεθνή προστασία ενηλίκων ε, σε καθένα από τα κράτη-μέλη. Σημαντική όμως διάκριση πρέπει να κάνουμε μόνο προς το εξή. Τα κράτη-μέλη που δεν είναι συμβαλόμενα στη Σύμβαση της Χάγης φαίνεται να παρουσιάζουν μια κατάσταση πολύ πιο δυσάρεστη, πολύ λιγότερο ικανοποιητική δηλαδή σε γενικού όρου. Ενώ εκείνα που έχουν κυρώσει τη σύμβαση μπορεί να έχουν κάποιε δυσκολίε, μόνο όμω στο μίσο που χρειάζεται συνεργασία με χώρε οι οποίε ακόμη δεν έχουν καταστεί συμβαλόμενα μέρη σύμβαση τη Χάγη. Οι δυσκολίε είναι τέτοιε που οι αρχέ των πρώτων κρατών ε, δεν μπορούν να αναπτύξουν πλήρω τα πλεονεκτήματα τις συμβάσεις θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας ενήλικας λοιπόν που ζει στη Γαλλία, ας πούμε ότι χέρι του ε, μέτρου προστασίας από δικαστήριο της Γαλλίας με κάποιον ε, που έχει επιφορτιστεί με την προστασία του ή την υποστήριξη του ε, πρώτου σε σχέση με τα οικονομικά και προσωπικά του συμφέροντα. Ο επιμελητής αυτός λοιπόν αναγκάζεται να μετακινηθεί σε κάποια άλλη χώρα. Σε μια χώρα που έχει ενδεχομένως ε, κυρώσει, μπορεί όταν μετακινηθεί στην Αυστρία να συνεχίσει να υπάγεται στην νομοθεσία της Γαλλίας και με υποστήριξη από τις αρχές της Αυστρίας δυνάμει της ε, συμβάσεως και αντίστροφα μπορεί να χρειαστεί οι αρχές της Αυστρίας να λάβουν από τις γαλλικές αρχές αρρωγή ε, ε, εάν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Μπορεί ακόμη υπό τη σύμβαση να μετακυληθεί η ευθύνη στις αυστριακές αρχές εάν κάτι τέτοιο απαιτείται από τα συμφέροντα του ενδιαφερομένου, κάτι το οποίο όμως δεν θα ισχύσει αν ο ενδιαφερόμενος μετά το, μετακομίσει στην Ιταλία, το Βέλιο, κάποια άλλη χώρα που δεν έχει κυρώσει τη σύμβαση. Αντίστοιχα λοιπόν η προστασία των δικαιωμάτων του αδύναμου ενηλίκου θα πρέπει να περάσει από το χάρτη για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα άτομα με αναπηρίες που όμως δεν μπορούν να δώσουν αποτελεσματική προστασία. Η Σύμβαση για την Προστασία των Ελληνικών τη Χάγη θα μπορούσε να αναπτύξει ένα πλήρε δυναμικό ε, αντιμετωπίζοντας έτσι τα κύρια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των ευάλωτων ενηλίκων σε περιπτώσεις διαμεθοριακές και ιδιαίτερα αυτό θα σημαίνει βελτίωση των συνθήκων σε όλη την Ευρώπη εφόσον ε, οι λύσει που περιλαμβάνονται σε αυτή τη σύμβαση γίνονταν κοινό αγαθό και κτήμα όλων των κρατών. Δύο τρόποι υπάρχουν λοιπόν για ένα πανευρωπαϊκό ε, καθεστώς ε, για την προστασία των αδύναμων ελίκων σε περιπτώσεις υπερσυνοριακές που αναφέρει η συνθήκη της Χάγης. Η πρώτη επιλογή έχει να κάνει με τα νομοθετικά μέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμει του άρθρου 80 τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα μπορούσαν να αντλήσουν έμπνευση και ίσω και κάποιε συγκεκριμένε διατάξει από την Σύμβαση τη Χάγη. Η δεύτερη λύση θα ήταν ε, ω εξωτερική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καλέσει η Ένωση τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ακόμη κυράσει, κυρώσει τη Σύμβαση της Χάγης ή προσχωρήσει σε αυτήν να το πράξουν προς το συμφέρον της Ένωσης με συνδυασμό των άρθρων 81 και 116 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί πιστεύουμε ότι η Ένωση δεν μπορεί να, πραγμα... δεν μπορεί να ε, καταστεί συμβαλόμενο μέρο συνθήκη τη Χάγη, καθώ αυτή είναι ανοιχτή σε συμμετοχή μόνο σε κυρίαρχα κράτη και όχι σε ε, πολυεθνικού οργανισμού. Η εξωτερική αρμοδιότητα πάντω τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλύση θα έπρεπε να προτιμηθεί για έχει περισσότερα πλεονεκτήματα, γιατί αυτό σημαίνει ένα δεσμευτικό νομικό εργαλείο και νομοθέτημα που θα, που θα δεσμεύει τα ε, κράτη-μέλη αλλά και τρίτα κράτη και θα οδηγεί σε μια οικουμενική αντιμετώπιση των ε, ζητημάτων κατά τον ίδιο τρόπο και ομοιόμορφη αξιοποίηση των ωφελημάτων της Σύμβασης της Χάγης για όλα τα κράτη-μέλη και αντίστοιχα και σε για χώρες μη ευρωπαϊκές που θα δεσμεύονται επίσης από τη Σύμβαση. Πρόκειται για μια προσέγγιση την οποία έχουμε δει και σε σχέση με τη Σύμβαση της Χάγης του 1996 για την προστασία των παιδιών που αυτή τη στιγμή είναι δίκαιο που δεσμεύει όλα τα κράτη-μέλη και πέραν αυτών. Πάντω, εάν προτιμηθεί η πρώτη λύση, ευρωπαϊκά νομοθετικά μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο το πεδίο της ε, προστασίας της Σύμβαση της Χάγη για τους ε, ανίκανους ή αδύναμους ενηλίκους, θα μπορούσαν να είναι μια λύση με συμπληρωματική ε, κάλυψη από τη Σύμβαση της Χάγης ε, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν από την ε, νομοθεσία την ευρωπαϊκή κάποιες αδυναμίες της Σύμβασης της Χάγης. Η μελέτη μας εντοπίζει πέντε πιθανές δυνατότητες βελτίωσης του νομοθετικού κειμένου της Σύμβασης της Χάγης σε περίπτωση που η λύση για, μια, ομοιόμορφη, για έναν ομοιόμορφο νομικό καθεστώς επιλεγεί και εισαχθεί αντίστοιχο νομοθέτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα θα προτείναμε τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού πλήρε εξουσίου για την προστασία ενηλίκου με απλούστευση της ε, παρουσίασης αποδεικτικών στοιχείων ως προς την ύπαρξη ε, και το περιεχόμενο ως εξουσίου για ε, ανήλικο υποπημέλεια. και σχετικά πληρεξούσια. Υπάρχουν διαφορές λοιπόν και για το κληρονομητήριο που θα μπορούσαν να καλυφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο από ένα γενικό πιστοποιητικό. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα για τον ανήλικα ανάλογα με το δίκαιο το οποίο επιλέγει να προσδιορίζει ε, την ένωμη τάξη του κράτους δικαίου του οποίου τα δικαστήρια θα εφαρμόσουν τις συνθήκες που προβλέπει η Σύμβαση της Χάγης για την προστασία του ανάλογα βέβαια και με το δίκαιο το οποίο καλύπτει το συγκεκριμένο πληρεξούσιο και πολύ συγκεκριμένα μπορώ να σας δώσω πτυχές της ερευνάς, σας, μας αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζωέλ Λόγκ έχει τώρα το λόγο. Όχι. Όχι, ευχαριστώ. Νομίζω κάλυψε και αυτά που θα είχα να πω εγώ ο καθηγητής ε, Μπριζίνα. Ωραία, τότε η κυρία Περζέγον για να κλείσουμε θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω θερμά τους δύο ε, ομιλητές οι οποίοι ε, σκιαγράφησαν πολύ καλά το θέμα. Βέβαια 15%, 15 λεπτά δεν φτάνουν να καλύψουμε ε, το θέμα των ευάλωτων ανηλίκων. 35% πάνω από 60% και έχουμε και πολλούς πάνω από 90%. Σε ό,τι αφορά την προστασία των ευπαθών ε, ενηλίκων δεν έχουμε πολλά. Ε, Παρόλα αυτά δεν πρόκειται για πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Έχουν δικαίωμα, είναι ίσα απέναντι στον νόμο και έχουν και αυτό δικαίωμα να μετακινούνται στην Ευρώπη. Είναι λοιπόν κατεπήγον και χρήσιμο να υπάρξει και σχετική νομοθεσία για αυτούς. Δεν θέλω να επανέλθω σε όλα όσα υπόθηκαν, διότι οι ειδικοί σχεγράφησαν πάρα πολύ καλά τα όλα προβλήματα. Μίλησαν για τη σύμβαση της Χάγης, που πράγματι είναι ένα εργαλείο, πολύ καλό νομοθετικό εργαλείο, το οποίο όμως δεν έχει επικυρωθεί από πολλές χώρες. Επομένως, δεν μπορεί και να εφαρμοστεί στην πράξη και δεν καταλαβαίνω γιατί η νομοθεσία ε, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα ήταν κάτι που δεν θα ήταν σκόπιμο. Εγώ πιστεύω ότι αντίθετα μπορούμε τι ανδρές γραμμές της μας Χάγης να ε, τις ε, συμπεριλάβουμε σε μια ευρωπαϊκή νομική πράξη. Βέβαια υπάρχουν πράγματα τα οποία λείπουν το ευρωπαϊκό πιστοπτικό για παράδειγμα με το οποίο δίνεται καθεστώς ευπαθού ή ευάλωτου ενηλίκου σε ένα άτομο χωρίς να πρέπει να ξαναρχίσει όλη διαδικασία όταν αλλάζει χώρα. Ε, για να ξαναχαρακτηριστεί ως ευάλωτος ενήλικος. Ξέρετε ότι ένας ευάλωτος, ένας ευπαθής ενήλικος ε, δεν μπορεί να συνάψει σύμβαση ε, ή συμβόλο που μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό και αναγκαίο για την καθημερινή του ζωή και θα πρέπει να τον συναντεύει κάποιος άλλος, αυτός που έχει το πληρεξούσιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Όλοι ίσως χρειαστούμε κάποια μέρα αυτή την προστασία Καλό είναι αυτό βέβαια και το εύχομαι γιατί σημαίνει ότι θα έχουμε φτάσει σε βαθιά γυρατιά όλοι μας και μακάρι να ζήσουμε πάρα πολλά χρόνια όλοι μας αλλά παραλαμβάνω πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα πρέπει να καταλάβουμε ότι αφορά ε, το μέλλον των ηλικιωμένων και ατόμων που έχουν κάποια αναπηρία, που βρίσκονται σε αδυναμία, ε, μπορεί να ε, πλήττονται και από ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας, ένα ψυχιατρικό πρόβλημα είναι λοιπόν σημαντικά όλα αυτά. Ε, καλό θα ήταν πιστεύω να δηλώσουμε ότι είμαστε υπέρ μιας ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Γιατί να μην υπάρχει. Ε, υπάρχουν και κάποιοι ε, που υποστηρίζουν την εθνική κυριαρχία, δεν τους βλέπω εδώ. Μα δεν θέλουμε να αλλάξουμε τα συστήματα και Απλά θέλουμε να αναγνωρίσουμε ένα ευρωπαϊκό καθεστώς ατόμων ευάλωτων, ενηλίκων ευπαθών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Κάστερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να στρέψω τη συζήτηση σε μια άλλη πτυχή. Έχουμε το πρόβλημα της γέρανσης του πληθυσμού και βλέπουμε ότι υπάρχουν ηλικιωμένοι, πολύ ηλικιωμένοι και το ποσοστό τους ε, θα αυξηθεί. Μιλάμε για τη λεγόμενη τέταρτη ηλικία και αυτή είναι η πλέον ευπαθής και για αυτή την τέταρτη ηλικία στην Ευρώπη θα πρέπει να ορίσουμε πολύ ξεκάθαρα διάφορες ε, συνθήκες πλαίσιο, παραδείγματος χάρη για την ε, ε, μέρημνα, την περίθαλψη των ατόμων αυτών για να μπορούν να ζουν αξιοπρεπώς. Είπαμε επίσης ότι θέλουμε να ενθαρρύνουμε την κινητικότητα μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι περισσότεροι ενήλικοι που χρειάζονται φροντίδα είναι ηλικιωμένοι και θέλουν να έχουν αυτή τη φροντίδα μέσα στο, ε, στην οικογένειά τους. Άρα τα μέλη της οικογένειας είναι οι φροντιστές στις περισσότερες περιπτώσεις. αυτό θα πρέπει να βρούμε κάποιες νομικές λύσεις και να υπερκεράσουμε τα προβλήματα που τίθενται. Στη Γερμανία αυτή τη στιγμή συζητούμε αυτό το ζήτημα και μας απασχολεί το κατά πόσον και σε ποιο βαθμό δεν υπάρχει και ένα είδος οργανωμένου εγκλήματος ε, που έχει να κάνει με τη φροντίδα στο σπίτι. Παίρνουν ε, χρήματα κάποια και από τα ταμεία υγείας. Αλλά δεν παρέχουν καμία φροντίδα. Άρα τίθεται στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι μπορεί να γίνει για να διατηρήσουμε ε, τις υπηρεσίες φροντίδας και κατοίκων φροντίδας σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Πρέπει επίσης να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ της διατήρησης ε, καλού βιωτικού επίπεδου και του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής. Γιατί όταν παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες φροντίδας ε, κατοίκων, οι αρχές θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση αλλά χωρίς και να παρεμβαίνουν ε, στις ε, λεπτομέρειες της ιδιωτικής ζωής κανενός. Είναι λεπτό το όλο θέμα, αλλά το σημαντικό είναι να μπορεί να ζει ένας ηλικιωμένος αξιοπρεπός. Ευχαριστώ. Κάποιος από τους ε, προσκεκλημένους μας θέλει να απαντήσει στις ερωτήσεις. Um... Δεν θέλω ακριβώ να απαντήσω σε αυτές τις παρατηρήσεις, απλώς θα ήθελα να διευκρινίσω μία πτυχή. Υπάρχουν διάφορα θέματα γύρω από την προστασία των ανηλικών, ευπαθών ανηλίκων και ένα από αυτά είναι η βοήθεια ή οι δραστηριότητες από ιδιωτικές ή δημόσιες αρχές για να φροντίσουν το άτομο αυτό. Η μελέτη μας αφορά όμω κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι οι πτυχέ του ιδιωτικού δικαίου που εμπλέκονται στο θέμα της προστασίας των ενηλίκων. Δηλαδή, ποιο δικαστήριο έχει δικαιοδοσία για να αξιολογήσει εάν ο ενήλικας αυτός ε, έχει πρόβλημα δικαιοπραξίας. Ε, τι μέτρα προστασίας θα πρέπει να δοθούν στο συγκεκριμένο άτομο. Δηλαδή, ε, να του οριστεί κάποιος και δαιμόνας, με ποιο δίκαιο εκπροσωπείται το άτομο αυτό, Ποιο είναι ο άνθρωπος ο οποίος εκπροσωπεί τον, τον, τον εν λόγω ενήλικα σε περίπτωση που θέλει να αγοράσει ή να πουλήσει ένα αγαθό κτλ. κτλ. Δηλαδή υπάρχουν διάφορες πτυχές ε, που έχουν να κάνουν την προστασία των ενηλίκων, αλλά όταν εμείς μιλούμε για την προστασία των ευπαθών ενηλίκων υπό τη Σύμβαση της Χάγης εστιάζουμε στο ιδιωτικό δίκαιο, που είναι μία από τις πτυχές που αφορούν την, ε, τα θέματα του ευπαθούς ανηλίκου. Ευχαριστώ. Και να προσθέσω και εγώ κάτι σε αυτό. Το άκουσα από δύο ευρωβουλευτές. Ένα από τα βασικά θέματα τα οποία έχουν προκύψει για τους ευπαθείς ή είναι ότι φυσικά ο ευπαθής ενήλικας ε, είναι κάτι πιο ευρύ από τον ευπαθή ηλικιωμένο. Δηλαδή, από τη στιγμή που ενηλικιώνεται κανεί, οποιοδήποτε ο οποίο ε, έχει κάποιο πρόβλημα, α πούμε, ένα 20χρονο μπορεί να έχει ένα ατύχημα και κάτι να του συμβεί και να έχει λοιπόν ανικανότητα δικαιοπραξία. Όλοι αυτοί οι ενήλικες εμπίπτουν στο πεδίο ε, της προστασίας. Η αρχική σύμβαση και οι αρχικές προτάσεις απορρέουν φυσικά από την αυξανόμενη κινητικότητα και από την γύρωση του πληθυσμού. Άρα καλύπτεται όλος ο πληθυσμός εκεί που μπορεί να έχει πρόβλημα και να χρήζει προστασίας. Σας ευχαριστώ όλους όσους ήρθατε να μιλήσετε για αυτό το θέμα. Ελπίζω να σας ξαναδώ στο μέλλον. Και θα συνεχίσουμε τώρα με ένα άλλο σημείο που είναι η ακρόαση για τον εξυγχρονισμό των κανόνων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα πνευματικά δικαιώματα. Το θέμα της φορητότητας όλος ιδιαίτερος θα συζητήσουμε. Okay, uh, Κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε. Έχουμε μείνει και πίσω στην ημερήσια διάταξη. Θα σας παρακαλέσω να συνεχίσετε τα πηγαδάκια εκτός εθούσης, παρακαλώ. Να κινήσω Καλωσορίζοντας καταρχάς ε, τους ε, προσκεκλημένους μας ε, στη δημόσια αυτή ακρόαση για τον εξυγχρονισμό των κανόνων περί δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτήτας και δι για τα θέματα αφορητότητας. Επίκαιρο το θέμα. Ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις κατέθεσε σχετική πρόταση και η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Η Επιτροπή Γιούρη είναι καθήλυνα αρμόδια για το Κοινοβούλιο. Υπάρχουν και δύο ακόμη, ΙΜΚΟ, ΚΑΛΤΑ, που θα είναι οι συνδεδεμένες επιτροπές στο πλαίσιο της όλης συζήτησης. Δεν έχω άλλες παρατηρήσεις, οπότε θεωρώ ότι μπορούμε να περάσουμε στις παρουσιάσεις από τους εμπειρογνώμονες. η κυρία Μαρία Μάρτιν Πράτ από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Connect. Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η πρώτη που θα λάβει το λόγο, παρακαλώ. Και να πω ότι σας ε, παραχωρώ 10 λεπτά στον καθένα, το πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είπατε κι εσείς ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 9 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα πέρυσι, δηλαδή ενέκρινε μια πρόταση κανονισμού για τη διευκόλυνση της φορητότητας των υπηρεσιών επιδραμικού περιεχομένου. Είναι ένα μέτρο που εντάσσεται ε, στη δέσμη πρωτοβουλειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο τη διευκόλυνση της λειτουργίας της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Στόχος όπως άλλωστε φαίνεται ξεκάθαρα και από τον τίτλο τη πρότασης είναι η εξασφάλιση της διασυνοριακή φορητότητα ε, των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου. Σε αυτή τη χρονική στιγμή θεωρώ ότι είναι σημαντικό να επιμείνουμε στον στόχο ότι δηλαδή ο στόχος είναι η διασυνοριακή φορητότητα. Δεν είναι ε, κάτι περισσότερο από αυτό. Με άλλα λόγια, η πρόταση δεν αποσκοπεί στην εξασφάλιση της δύο συνεργικής πρόσβασης υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται σε κράτος μέλος, το οποίο είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος συνήθως διαμονής ε, του καταναλωτή. Και γιατί επιμένουμε σε αυτό ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιμένουμε διότι όπως γνωρίζετε είχαμε τις συζητήσεις για την εδαφικότητα και το πώς επηρεάζει τον κλάδο ε, το σχετικό και στην ανακοίνωση της DSM του Μαΐου και είχαμε και την ε, ανακοίνωση ε, για το copyright και όλα αυτά πιστεύω ότι ξεκαθαρίζουν ότι θέλουμε μια βαθμιδόν προσέγγιση και κάνουμε το πρώτο βήμα ακριβώς με αυτή την ε, ανακοίνωση για την φορητότητα. Είναι μια στοχευμένη πρόταση και φιλόδοξη πρόταση ταυτόχρονα ε, είναι μια πλήρης, μια περιεκτική πρόταση για την ενιαία αγορά. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι είναι και μια πρόταση που ξεπερνάει το, τα δικαιώματα δημιουργού, το copyright. Έχουμε έναν ορισμό για τις επιγραμμικές υπηρεσίες στον κανονισμό. Αυτός ο ορισμός καλύπτει όλες τις υπηρεσίες επιγραμμικού περιεχομένου και όχι μόνο τις υπηρεσίες που ε, παρέχουν ε, πρόσβαση σε περιεχόμενο προστατευμένο από τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας. Είχαμε και τα σχετικά με τους κατόχους δικαιωμάτων σε αθλητικές διοργανώσεις. Υπερβαίνει το copyright γιατί δεν θεσπίζει απλά κανόνες που είναι σημαντικοί σε ό,τι αφορά τον ορισμό και την άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής διοκτησίας, αλλά αφορά και τους παρόχους υπηρεσιών, επιβάλλει υποχρεώσεις στους παρόχους υπηρεσιών και θα επανέλθω στο θέμα αυτό όταν θα διατρέξω τα άρθρα της πρότασης εν συντομία. Όπως είπα, το πεδίο εφαρμογή είναι επιγραμμικές ε, υπηρεσίες, υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου που παρέχονται νομίμως. Αυτό είναι σημαντικό. Βλέπετε τα σχετικά στους ορισμούς της πρότασης ε, κανονισμού. Μιλούμε δηλαδή πραγματικά για υπηρεσίες ε, που είναι κεκριμένες, ε, έχουν εγκριθεί από τον κάτοχο δικαιωμάτων και παρέχονται στους καταναλωτές σε φορητή βάση στη χώρα διαμονής, συνήθως διαμονής του καταναλωτού. Θέλουμε δηλαδή η φορητότητα να γίνεται και διασυνοριακά. Στόχος του κανονισμού πάνω απ' όλα είναι να καλύψει τις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται έναντι αμοιβή, ε, έναντι καταβολής μετρητών από τον ε, καταναλωτή. Συνδρομητικές τις λέμε είναι σε αυτές τις υπηρεσίες ε, και υπάρχει η δυνατότητα, έτσι προβλέπεται στο κείμενο και θέλουμε να ξεκαθαριστούν οι σχετικές αμφιβολίες και απόρριες που υπάρχουν. Ό,τι λοιπόν αναφέρεται υπάρχει αυτή η δυνατότητα στο κείμενο γιατί και οι πάροχοι υπηρεσιών να καλύπτονται και εφόσον δεν παρέχουν υπηρεσίες εναντί ε, πληρωμής, υπάρχουν σκαρδία, φήμηση ή μπορεί να καταβάλουν ένα τέλος ε, τηλεοπτικών δικαιωμάτων κτλ. Δεν καλύπτονται αυτόματα όλα αυτά. Η πρόταση εστιάζει σε δύο πυλώνες κυρίως. Υπάρχει ένα νομικό πλάσμα, ένα legal fiction που λέει που λέει ότι πρόσβαση υπηρεσίες από τον καταναλωτή υποτίθεται ότι θα γίνεται πάντοτε στην χώρα συνήθως διαμονής ακόμη και όταν ο καταναλωτή καταναλωτής έχει πρόσβαση στην υπηρεσία επιγραμμικού περιεχομένου εκτός της χώρας της διαμονής του. Με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό γίνεται σε προσωρινή βάση. Και με αυτό το νομικό πλάσμα ουσιαστικά βοηθούνται οι πάροχοι των υπηρεσιών για να είναι σαφή τα δικαιώματα. Όταν οι συνδρομητές δηλαδή είναι εκτός του χώρου συνήθω διαμονίζουν για κάποια περίοδο σε κάποια άλλη χώρα τη Ένωση να μπορούν να έχουν εξασφαλισμένο αυτό το δικαίωμα. Δεύτερη σημαντική πρόταση είναι η υποχρέωση ε, εξασφάλιση τη φορητότητα. Η υποχρέωση τους, ε, στου παρόχου να την εξασφαλίζουν τη φορητότητα. Στο άρθρο 3 προβλέπεται αυτό. Λέμε δηλαδή στους παρόχους υπηρεσιών ότι πρέπει να εξασφαλίσουν τη φορητότητα, έχουν τη σχετική υποχρέωση. Μέχρι στιγμή δεν υπήρχε αυτή η υποχρέωση να εξασφαλίσει ο πάροχος υπηρεσιών την ίδια ποιότητα της υπηρεσίας όταν ο καταναλωτής δεν ε, βρίσκεται στη χώρα διαμονής, στο είδος διαμονής. Υπάρχει και ένας άλλος νοτερισμός, μια άλλη καινοτομία στην όμθεση αυτή. Υπάρχει ένα άρθρο, το άρθρο 5 συγκεκριμένα, το οποίο βασικά εξασφαλίζει το ότι δεν μπορεί να παρακάμψει κανείς την υποχρέωση που θεσπίζεται από τον κανονισμό με, συμβατική, με κάποιο συμβατικό διακανονισμό η διευθέτηση. Είπα και στην αρχή της παρέμβασής μου ότι πρόκειται για μια περιεκτική ε, διεξοδική νομική πράξη που αφορά την εσωτερική αγορά. Βέβαια βλέπετε ότι ε, επειδή είναι κανονισμός, υπάρχει και η δυσκολία το ότι θα πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρος ο κανονισμό να μπορεί να εφαρμοστεί μετά. Πρέπει να είναι όλα πάρα πολύ ε, σαφή λοιπόν μέχρι να τεθεί σε ισχύ αυτό το νομικό μέσο. Ένα νομικό μέσο που θα είναι άμεσα εφαρμοστέο στην αγορά και σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μεταξύ ιδιωτικών ε, συμβαλωμένων, ιδιωτικών φορέων. Άρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι από τη μία Θέλουμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή προβλεψιμότητα και σαφήνεια για την αγορά. Και από την άλλη πλευρά, όπως συμβαίνει πάντοτε όταν ρυθμίζουμε ένα τομέα που έχει να κάνει με τεχνολογίες, θέλουμε να καταλήξουμε σε λύσεις που θα είναι στο δυνατόν αξιόπιστες. Επαλήθευση ποιοι είναι οι μηχανισμοί επαλήθευση που θα πρέπει ε, να έχουμε για να μπορούμε να τεκμηριώνουμε ποια είναι και η χώρα συνήθω διαμονή ε, του ε, καταναλωτή. Η Προεδρία του Συμβουλίου έχει καταβάλει σημαντικέ προσπάθειε, έχει εστιάσει σημαντικά σε αυτή την πρόταση και πρέπει να σα πω ότι όταν συζητούμε με τα κράτη-μέλη τη σχετική αυτή πρόταση, συχνά ε, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι έχουμε ένα τρίγωνο. Έχουμε τη διαμονή, την πρώτη κατοικία, έχουμε δεύτερο, δεύτερη γωνία τα μέσα επαλήθευσης και το τρίτο, η τρίτη γωνία του τριγώνου είναι η προσωρινή διαμονή. Και οι προσπάθειές μας πρέπει να εστιάσουν στην όσο το δυνατόν πιο σαφή διευκρίνηση, στον πιο σαφή ορισμό της αρχής αυτής, του ορισμού της έννοιας ε, πρώτη ή συνήθις διαμονή και πώς μπορεί αυτή να επαληθευτεί. Αυτά τα δύο στοιχεία νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσουν περισσότερο και όχι τόσο το να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε τη φορητότητα. για κάποιον ο οποίος προσωρινά διαμένει κάπου αλλού. Μιλάμε για τη φορητότητα στην εσωτερική αγορά υπηρεσιών για τι οποίε έχει πληρώσει ο καταναλωτή. Έτσι σα το υπενθυμίζω. Δεν μιλάμε για ε, υπηρεσίε που δεν έχει πληρώσει ο καταναλωτή, ούτε μιλάμε για κάτι που σημαίνει ζημία προ τον κάτοχο του δικαιώματο. Απλά λέμε ότι ένα καταναλωτή που έχει πληρώσει για κάποιε υπηρεσίε στην συνήθι ε, κατοικία του, συνήθι τόπο διαμονή του, να μπορεί να απολαμβάνει των υπηρεσιών αυτών να προσωρινά διαμείνει κάπου αλλού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρόζενμπεργκ είναι ο επόμενος ομιλητής, που είναι επικεφαλής του τμήματος Engineering στη Sky. Ε, θα ακούσουμε την προσέγγιση, την τεχνική του θέματος. Λέγομαι Ρίτσαρντ Ρόζενμπεργκ. Έχετε 10 λεφτά, λέει ο πρόεδρος. Δουλεύω εδώ και 20 χρόνια σε αυτόν τον τομέα της τεχνολογίας, τελευταία 15 στο Sky Είμαι αρχιμηχανικός, είμαι υπεύθυνο από την αρχή όταν δημιουργήσαμε το Sky, ε, τις τηλεοπτικές υπηρεσίες ε, online το 2011 ασχολούμαι με αυτά. Θέλω αυτά τα 10 λεπτά που έχω να μιλήσω για τις τεχνικές δυσκολίες, ε, φυσικά για διασυνοριακή φορητότητα. Θα ήθελα να κάνω μια εισαγωγή στο Sky όμως, ποιες είναι οι αξίες μας, ποιες είναι οι αρχές, και πώς βλέπουμε την φορητότητα. Είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία ψυχαγωγίας, ε, συμβάλλει στην ευρωπαϊκή οικονομία, 10 ε, δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στον ευρωπαϊκό ΑΕΠ. Έχουμε 21 εκατομμύρια πελάτες σε 5 χώρες. Είμαστε στην Ιταλία, Γερμανία, Αυστρία, Ιρλανδία και φυσικά στο Μενοβασίλειο. Πάνω απ' όλα, Είμαστε μια αισιόδοξη εταιρεία, πιστεύουμε ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι και θέλουμε να έχουμε το καλύτερο περιεχόμενο, την μεγαλύτερη ε, καινοτομία, τις καλύτερες υπηρεσίες για τους πελάτες. Ε, εξοδεύουμε 7 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε όλη τον όμιλο και ξέρετε πολύ καλά ότι δίνουμε και παρέχουμε και αθλητικές, αθλητικό θέαμα, ε, ταινίε κτλ. Αλλά έχουμε και δικά μας θέαματα, μεγάλα shows όπως τον Κομόρα και το Fortitude. Αυτές είναι, αυτά είναι κάποια από τα show που ε, δίνουμε. Θέλουμε να είναι πολύ καλό το περιεχόμενο που δίνουμε στους πελάτες μας, με ένα απλό τρόπο. Ε, και έχουμε και μια υπηρεσία, είμαστε πρώτη στις ε, υπηρεσίες ε, περιεχομένου. Ε, εξοδεύουμε 400 εκατομμύρια για τη βελτίωση του, του περιεχομένου που δίνουμε στους πελάτες μας μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, για την διασυνοριακή φορητότητα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εξέλιξη. Θέλουμε να την προσφέρουμε στους πελάτες μας που ό,τι κάνουμε το κάνουμε για αυτούς. Το βασικό είναι ότι Χρειάζεται όμως προσπάθεια για να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά την αρχή αυτή, γιατί θα πρέπει να είναι και απλή και να είναι εύχρηστη για τους πελάτες, χωρίς να υποσκάψουμε την εδαφική αποκλειστικότητα που έχουμε με βάση τις συμβάσεις μας. Βασιζόμαστε λοιπόν στις εξής τρεις αρχές. Πρώτον, θέλουμε να επαληθεύσουμε ότι οι πελάτες τους οποίους δίνουμε τη φορητότητα είναι πραγματικοί πελάτες, χωρίς όμως να εισβάλλουμε στην ιδιωτική του σφαίρα. Πέρα από τις νομοθετικές υποχρεώσεις υπάρχει και μια ηθική, δηλαδή η εμπιστοσύνη των πελατών μας μας ενδιαφέρει τα μάλλα. Δεύτερον, ανταγωνιζόμαστε για τις βασικές μας υπηρεσίες, τις καλύτερες, με, την, με το Netflix και το Amazon, με τους άλλους μεγάλους παίκτες. Επομένως, οι έλεγχοι θα πρέπει να είναι αποτελεσματικοί, αλλά όχι να μας βάζουν σε μειονεκτική θέση και να μην ε, είναι πολύ επαχθεί για τους πελάτε. Θα πρέπει να είναι απλή για τους πελάτε μας. Και τέλος, δεν θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ένα απλό προϊόν και να εξασφαλίσουμε την φορητότητα εγκαίρω, εάν θα πρέπει να διαπραγματευόμαστε ειδικού όρου με κάθε ένα από τους 700 ε, ε, προμηθευτές περιεχομένου με τους οποίου συνεργαζόμαστε. Τώρα, να πάμε στις τεχνικές και επιχειριακές ε, δυσκολίες και προκλήσεις. Όπως είπα και προηγουμένως, η διαδικασία εφαρμογή της φορητότητας είναι πάρα πολύ περίπλοκη και δεν θα πρέπει να υποτιμήσουμε τη δυσκολία. Έχουμε ε, διάφορες υπηρεσίες ε, σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές και οι τεχνικές πλατφόρμες που υποστηρίζουν την παροχή αυτών των υπηρεσιών δημιουργούνται με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να υπάρχει συμβατότητα με ένα ευρύ, μια ευρύ φάσμα πούμε, τρίτων φορέων. Ας πούμε. Έχουμε λοιπόν λογισμικό σε ταμπλέτες, σε κινητά, ε, σε κονσόλες παιχνιδιών, σε επιτραπέζους ε, υπολογιστές κτλ. κτλ. Και όλο αυτό το πολλαπλό, ας πούμε, αυτό το πλέγμα αυτό τον, του λογισμικού έχει διάφορες ε, λειτουργικές, ας πούμε, παραμέτρους, έτσι. Κάθε, φορά που ένας κατασκευαστής αναβαθμίζει, ας πούμε, την εφαρμογή στο, εμείς θα πρέπει να ξαναδούμε το λογισμικό μας, που ώστε να μπορεί να λειτουργεί. Επομένως, πρέπει να εξετάσουμε τις επιπτώσεις της φορητότητας και αυτό κάνουμε τώρα. Το βασικό όμω είναι ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να γίνει ε, σε όλο το λογισμικό μας και αυτή είναι μια πολύ ε, παχθή διαδικασία, δύσκολη και περίπλοκη. Δεύτερον, θέλουμε να δίνουμε ε, τέλειο, τέλεια ποιότητα ε, επιγραμμικού περιεχομένου βίντεο κτλ. στου πελάτε. Μπορώ να μιλάω για ώρε για αυτό το θέμα, με ενδιαφέρει πολύ. Αλλά η ποιότητα ενός, ε, μιας εκπομπής, ας πούμε, επιγραμμικά, το θέμα δεν είναι μόνο ο αριθμό των πιξελών, ε, δεν είναι μόνο το resolution, δεν είναι μόνο η ευκρίνεια δηλαδή, αλλά είναι και η εμπειρία που έχει ο πελάτης. Και αυτό θέλουμε συνεχώς να το βελτιώνουμε. Και εκεί ο Sky ε, επενδύει, δηλαδή έχουμε τη δική μας υποδομή, Ε, για τα μεμονωμένα ISP. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα των υπηρεσιών ε, θα πρέπει να καθορίζεται από την αγορά. Και αν ε, οι πελάτες θέλουν να βελτιώσουν την εμπειρία τους σε σχέση με το, με το τι βλέπουν, ας πούμε, όταν ταξιδεύουν στο εξωτερικό, θα πρέπει να τους λάβουμε υπόψη μας. Θα πρέπει να έχουμε καλέ πλατφόρμε καταρχά και είναι περίπλοκη διαδικασία αυτή όπω σα είπα, γιατί το, η ασφάλεια του περιεχομένου και των δεδομένων των προσωπικών του πελατών μα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μα. Πιστεύουμε ε, ότι θα πρέπει να ε, επαληθεύουμε αποτελεσματικά την κατοικία, θα πρέπει να βλέπουμε τι μεθόδου πληρωμή που χρησιμοποιούν οι πελάτε στην αρχική φάση συναψή του συμβολέου και συνεχεία ε, από μήνα σε μήνα και να συνδέεται με συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό στη χώρα κατοικία, Αλλά δεν αρκεί αυτό. Επίσης πιστεύουμε ότι οι συνεχεί ε, έλεγχοι χρειάζονται για να μην υπάρχουν ε, καταχρήσεις. Επίσης, χρήσιμο θα ήταν η νομοθεσία να μας επέτρεπε ένα πελάτης ο οποίος έχει μία υπηρεσία ε, αλλά ποτέ δεν τη χρησιμοποιεί στη χώρα κατοικία να ζητάμε από αυτόν επιπλέον αποδεικτικά στοιχεία για τη συνήθεια κατοικία. Τέταρτον, όσο ο κανονισμός επηρεάζει, μας επιβάλλει να επαληθεύουμε την κατοικία, ε, επομένω ε, προστατεύει ας πούμε, την εδαφική αποκλειστικότητα, δεν νομίζω ότι πρέπει να επιβάλλουμε χρονικού περιορισμού στου πελάτε μα. Ούτω ή άλλω προτιμούμε να μην το κάνουμε, καθότι δεν πιστεύουμε ότι θέλουν τέτοια όρια χρονικά και πιστεύουμε ότι είναι και πολύ περίπλοκο να του το εξηγήσουμε. Και τεχνικά για να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε ε, και να μην ενοχλούμε τους πελάτες θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και τέλος, ε, και σημαντικό, ε, η Κομισιόν κάνει νομοθετικές προτάσεις με στόχο τη μείωση των νομικών ασαφιών, ας πούμε, δημιουργώντας αυτό το νομικό πλάσμα που αναφέρθηκε και ο ε, πελάτης ε, να αισθάνεται στο κέντρο αυτής της ιστορίας, ανεξάρτητα από το που βρίσκεται σε ποια χώρα. Ε, ο ΣΚΑΙ καταλαβαίνει ότι δεν θέλουμε να ε, υπάρχουν τα, τα πνευματικά δικαιώματα παρά μόνο στο κράτος μέλος, μέλος που προβλέπεται. Νομίζουμε ότι ως νομικό πλάσμα είναι καλό, θα δίνει μεγαλύτερο περιεχόμενο στους ε, πελάτες, πιο γρήγορα από ό,τι αγορά, αλλά θα πρέπει ε, να εξασφαλίσουμε διάφορα πράγματα για να λειτουργήσει. Και θα πρέπει να είναι ευρύ. Επίσης, θα ήθελα να σας προτείνω κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να κάνουν οι νομοθέτες για να μας βοηθήσουν εμάς και άλλους Καταρχά έχουμε αυτές τις ε, λειτουργικές δυσκολίες. Αυτό το νομικό πλάσμα, όπως σας είπα, ε, μόρφωμα, ας πούμε, θα πρέπει να οριστεί ευρέω. καθόλου εξαιρέσει, καμία εξαίρεση να μην επιτρέπεται. Δεύτερον, η διαδικασία της επαλήθευση θα πρέπει να είναι αποτελεσματική και νομικά υποχρεωτική. Τρίτον, ε, η προσωρινή παρουσία. Δεν θα νομίζω ότι χρειάζεται χρονικός περιορισμός αν υπάρχει μια αποτελεσματική επαλήθευση, δεν χρειάζεται ε, χρονικό περιορισμό. Και σε ό,τι αφορά τη μεταβατική περίοδο, δεδομένων των ε, λειτουργικών δυσκολιών και περιπλοκών για την εφαρμογή, προβλέπουμε, προτιμούμε μάλλον ε, έξι μήνες μετά την υιοθέτηση του κανονισμού να έχουμε μια μεταβατική περίοδο όπου θα είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουμε αυτό το νομικό μόρφωμα, πούμε, αλλά όχι υποχρεωτικά στο τέλο της μεταβατικής περίοδου θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τη φορητότητα. Αυτοί που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τη φορητότητα αυτές του 12 μήνες να μην τιμωρούνται παρακαλώ. Αυτά, ευχαριστώ και είμαι έτοιμος να ακούσω και ερωτήσει μετά. Uh, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Αγκουστίν Ρέινα, Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών για να μας φωτίσει στην προοπτική των καταναλωτών. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι και ευχαριστώ και τη Γραμματεία για την πρόσκληση να τοποθετηθούμε. Ονομάζομαι Ρέινα, Αγκουστίν Ρέινα, εργαζομαι για την Οργάνωση Καταναλωτών της Ευρώπης, μια υπερεθνική οργάνωση των, ε, ένωση των οργανώσεων καταναλωτών που αγωνίζεται να τα δικαιώματα των καταναλωτών και να ενημερώνει για αυτά τους ε, αρμόδιους για τη λήψη των αποφάσεων. Ε, αναφέραμαστε λοιπόν στη μεταρρύθμιση του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας. Βεβαίως είναι πολύ ευρία η έννοια, τόσο είναι τα συμφέροντα αλληλοσυγκρουόμενα και πολλές φορές και σε αντίθεση με την ε, εθνική η νομοθεσία είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να συγκεράσει όλα ο νομοθέτης σε μία πρόταση. Από τη δική μου λοιπόν την προοπτική θα μιλήσω για τα δικαιώματα του καταναλωτή, για το πώς εμείς βλέπουμε την εξέλιξη αυτών των συζητήσεων για την νομοθεσία. Είναι πολύ καλό σημείο κίνησης ε, το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 9 Ιουλίου όπου το Κοινοβούλιο ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη διάσταση των καταναλωτών στη μελέτη των προτάσεων για, το, για την πνευματική ιδιοκτησία. Πρόκειται για την πρώτη φορά στην ιστορία όπου το Κοινοβούλιο επιμένει και εισάγει τη διάσταση του καταναλωτή για το δίκαιο της μηχανικής ιδιοκτησίας. Και έτσι η Επιτροπή καταθέτει την πρόταση που υπόθηκε νωρίτερα ότι έχει χαρακτηριστικά ιστορικής αγοράς θα συμπληρώσω εγώ χαρακτηριστικά δικαίου του καταναλωτή, δηλαδή η προσέγγιση, το μέλημα είναι η αντιμετώπιση, η πρόληψη, η θεραπεία των προβλημάτων που μπορεί να έχει ένας καταναλωτής να ταξιδεύει στο εξωτερικό και αγοράζει υπηρεσίες ή αγαθά. Ε, ένα μικρό βήμα λοιπόν μπορεί να είναι. Μικρό ναι γιατί, γιατί θα εξυπηρετήσει τον καταναλωτή εκείνον ο οποίος ταξιδεύει. Είναι όμως σημαντικό θα υπηρετήσει και τον καταναλωτή ο οποίος θα αγοράσει υπηρεσίες ε, στη χώρα, νομικές υπηρεσίες στη χώρα στην οποία ζει. Ε, και είναι σημαντικό λοιπόν ως βήμα διότι δείχνει πως το δικαίωμα της ιδιοκτησίας της πνευματικής, της μηχανικής αφορά και τον καταναλωτή και απαιτείται η διασφάλιση κανόνων δικαίου επακριβών, της ασφάλειας δικαίου δηλαδή και βέβαια, όπως είπε και η συνάδελφος νωρίτερα, τα ζητήματα της φορητότητας μπαίνουν σε αυτή την ε, προσέγγιση. Πώς λοιπόν θα αξιολογήσουμε την επιτυχία της πρότασης. Η Μαρία ήδη αναφέρθηκε στις διαφθορές πτυχές. Είναι πολύ απαραίτητο πιστεύω να υπάρχει ένα πεδίο, ένα, ε, μια θεώρηση ευρεία και ξεκάθαρη ε, της Σύμβαση καταρχά. Πρέπει να υπάρχει μια σύμβαση παροχή υπηρεσία, συνδρομής δηλαδή. Εφόσον υπάρχει σύμβαση πρέπει να υπάρχει και δυνατότητα φορητότητα. Άρα οι υπηρεσίε οι οποίε προσφέρονται χωρί να προηγείται σύμβαση αποκλείονται. Υπάρχει μια συζήτηση για το αν οι δωρεάν υπηρεσίε θα πρέπει να περιλαμβάνονται νέου. Εδώ ε, το κτηνητήριο ε, που μπήκε ήταν ε, τη ύπαρξη μια σύμβαση. Επίση δεν ορίζεται, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, χρονικό όριο για την φορητότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι μπορεί να έχει διαφορετικές ανάγκες φορητότητας ένας καταναλωτή. Μπορεί κανεί να ταξιδεύει για το εράσμο, για τη δουλειά του, για τι διακοπέ του. Διάφοροι λόγοι λοιπόν και αναλόγω δεν θα ήταν σκόπιμο να οριστεί ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο ε, ή συγκεκριμένο αριθμό εβδομάδων ή μηνών, επί παραδείγματι, που μπορεί κανεί να βρεθεί στο εξωτερικό. Πολύ θετικό επίση είναι το υποχρεωτικό, η υποχρεωτική διάσταση τη φορητότητα στον κανονισμό. Δεν μπορεί να περιοριστεί δηλαδή από διατάξει ιδιωτικού δικαίου, από συμβατικέ διατάξει και βάλιστα έχει και αναδρομική ε, λειτουργία. Αυτό σημαίνει ότι, δεδομένου μάλιστα ότι οι συμβάσει ε, είναι επιτοπλίστων μακροχρόνιε, ε, ε, θα ισχύσει και σε υφιστάμενε συμβάσει. Το πλάσμα δικαίου λοιπόν το που έχει εισαχθεί είναι μια πολύ καλή επιλογή για να ε, επιλεγεί ένα νομικό πλαίσιο ανάλογα με το κράτος μέλος. Τώρα το τι διευκρινίζεται η ανάγκη για την συνήθη κατοικία, διευκρίνηση της συνήθους κατοικίας, αναλογική και μη παρεμβατική για τον καταναλωτή είναι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ σωστά το επεσήμανε η συνάδελφος ο συνάδελφος του ΕΣΚΑΙ και επίσης θα πρέπει να προσφέρεται επαρκής ευελιξία για προσαρμογή στην ε, επιχείρηση. Είναι κανονισμός λοιπόν, πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη, ωστόσο θα έχει έναν μηχανισμό αξιοποίησης ο οποίος μπορεί για το μέλλον να δίνει λύσεις παρά τις όποιες εξελίξεις, αλλά ταυτόχρονα ίσως και θα πρέπει να επιμείνουμε στον τρόπο με τον οποίο θα υλοποιηθεί ο κανονισμός. Πάντως υπογραμμίζω ότι δεν είναι παρεμβατικός και κάνει σεβαστή την ιδιωτικότητα, τον ιδιωτικό βίο του καταναλωτή. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε, αν χρειάζεται, ότι συμβατικά δεν θα είναι αδύνατο να οριστούν ε, χρονικά όρια για τη φορητότητα. Υπάρχει δηλαδή υποχρέωση να χορηγηθεί η φορητότητα μέσα από τον κορονισμό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει και κάποιο παραθυράκι μέσα από το οποίο ένας ε, πάροχος θα μπορούσε να ε, επιβάλλει να εξασφαλίσει περιορισμό του χρονικό της φορητότητας. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί λοιπόν από την ε, περαιτέρω μελέτη. Επίσης η δυνατότητα ο καταναλωτής να έχει πρόσβαση σε ένα κατάλογο ε, τηλεφωνικό ο οποίος είναι διαθέσιμος σε κάποια άλλη χώρα. Για αυτόν ο οποίος ταξιδεύει συχνά. Πρόκειται για το ε, μάλλον για τον κατάλογο υπηρεσιών που προσφέρει ο πάροχος και σε ξένη χώρα. Για κάποιον που ταξιδεύει συχνά, αυτό είναι το φαινόμενο Netflix όπως το λέμε. Κάποιος που είναι σε μια χώρα εγκατεστημένος έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένο κατάλογο υπηρεσιών του Netflix, αλλά θα πρέπει, εάν ταξιδεύει και σε άλλη, να έχει δυνατότητα να συμβουλεύεται και άλλον κατάλογο και έτσι μπορεί να επιλέγει τον κατάλογο στον οποίο θέλει να έχει την πρόσβαση, δηλαδή το κατάλογο της χώρας της συνήθους διαμονής ή της χώρας στην οποία επισκέπτεται. Η τεχνολογική ουδετερότητα επίσης έχει πολύ σημαντική σημασία ως αρχή, ανεξαρτήτως δηλαδή του μηχανήματος που χρησιμοποιεί ο καταναλωτής πρέπει να έχει την ίδια πρόσβαση και η παρακολούθηση, επιτήρηση συγκεκριμένα της στήρησης των διατάξεων και της παράβασής τους. Για μας είναι πολύ καλή η πρόταση της Επιτροπής, είναι πολύ καλό βήμα. Καλούμε το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο να την υποστηρίξουν και να την υιοθετήσουν το ταχύτερο δυνατό, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στο επόμενο βήμα μια ευρύτερη μεταρρύθμιση. Και εδώ σε μία μόνο ε, διαφάνεια θα σας αναφέρω τι μπορούν να περιμένουν οι ενώσεις καταναλωτών ως επόμενο βήμα. Η Μαρία, η Μαρία ήδη το ανέφερε. Φορητότητα, προς το παρόν και μόνο φορητότητα, όχι δηλαδή υπερσυνοριακή πρόσβαση. Ε, την υπερσυνοριακή πρόσβαση θα την συζητήσουμε, ελπίζουμε, σε κάποια επόμενα ε, σύνολα μέτρων, σε κάποιες επόμενες προτάσεις, γιατί πιστεύουμε ότι και εκεί χρειάζεται παρέμβαση ρυθμιστική, κυρίως όσον αφορά την οδηγία για την ε, ε δορυφορική και καλωδιακή τηλεπικοινωνία. Επίσης υπάρχει οδηγία InfoShock, όπου μπορούν να υπάρχουν πολλές βελτιώσεις, πάντα έχοντας πως βεβαίως ότι μας περιορίζει ένα διεθνές πλαίσιο που ισχύει. Άρα δεν περιμένουμε τίποτε το υπαραστατικό. Υπάρχουν όμως σημαντικά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν από την οπτική γωνία του καταναλωτή, παρεκκλήσεις, περιορισμοί, αν χρειάζεται μία νέα παρέκκληση για περιεχόμενο παραγόμενο από τον χρήστη και άλλα τέτοια ζητήματα. Και για να ολοκληρώσω, η ΜΠΕΟΚ μαζί με άλλες ενώσεις έχει ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις θέσεις της σε σχέση με την επερχόμενη μεταρρύθμιση. Μια φιλόδοξη, πιστεύουμε, λύση ε, που ε, ενισχύει και τη δημιουργικότητα και την παραγωγή στην ερνή αγορά και τον καταναλωτή βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Σέσιλ Σπρίγκερ Εκτελεστική Διευθύντρια της ε, εταιρείας οπτικοακουστικής προσφοράς, ε, μάλλον παραγωγών οπτικοακουστικών παραγωγών, θα μας δώσετε και στις απόψεις. Ευχαριστώ. Για να μην βαρεθεί τα αγγλικά θα περάσω στα γαλλικά εγώ. Και δεν έχω και PowerPoint, άρα θα πρέπει να μ' ακούσετε απλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω που με επιλέξατε να σας εκφράσω την άποψη των δημιουργών. Η Ένωση των Δημιουργών Οπτικοακουστικού Περιεχομένου ε, είναι μία εταιρεία διαχείριση των δικαιωμάτων ε, των σκηνοθετών, σεναριογράφων ε, ε, και άλλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των οπτικακουστικών με 29 εταιρείε από 19 κράτη εκπροσωπούμε. Έχουμε προετοιμάσει κάποια σχόλια σε σχέση με την πρόταση κανονισμού της Κομισιόν. Στα αγγλικά έχω κάποια αντίγραφα μαζί μου, μπορώ να σας τα διαθέσω. Εγώ θα εστιάσω την ομιλία μου σε τέσσερα σημαντικά σημεία, διότι βέβαια δεν μπορώ μέσα σε 10 λεπτά να καλύψω όλο το φάσμα. Σίγουρα οκτώ άρθρα μόνο περιλαμβάνει ο κανονισμός, ωστόσο ε, γύρει πολύ σημαντικά ζητήματα, ζητήματα αρχής και ζητήματα πρακτικής φύσεως. Ε, ξεκινώντας από τα ζητήματα αρχής, ε, έχουμε λοιπόν επιτάπητος μια πρόταση κανονισμού, κάτι πρωτάκουστο για τον τομέα της νοματικής ιδιοκτησίας με στόχο τη δημιουργία υποχρέωσης διεσυνοριακής φορητότητας για τους κατόχους δικαιωμάτων, για τους δικαιούς, δηλαδή παρόχους υπηρεσιών μάλλον και δικαιούχων, ε, καταναλωτών συγκεκριμένα. Αυτή η υποχρέωση για τους δικαιούχους ξεκινά ε, μάλλον ουσιαστικά οδηγεί σε περιορισμό του δικαιώματος αν δεν μπορούν να φέρουν καμία ε, αντίσταση. Όπως είπε η Μαρία, έχουμε ένα πλάσμα δικαίου το οποίο προσθέτει, μάλλον προσδίδει κάποια δικαιώματα σε ό,τι αφορά και αναφέρεται στη συνήθεια κατοικία, στη διαμονή. Έχουμε περιορισμό και των κατόχων δικαιωμάτων και των δημιουργών, αλλά επίσης αντιβαίνει και στην αρχή της ενταφικότητας για τη χρήση των ε, διαφόρων έργων που κανονικά θα έπρεπε να ε, συνεπάγεται την κατοχή μιας πολύ ε, πολυεθνικής διασυνοριακής από πολιτικής πλευράς η δημιουργή δεν είναι αντίθετη στην ε, εφαρμογή μιας διασυνοριακής φορητότητας για να ληφθούν υπόψη εξελίξεις ε, στη χρήση και η ευρωπαϊκή κινητικότητα, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει ε, με βάση συγκεκριμένου όρου και την αυστηρή του εφαρμογή. Πρώτο όρο, πρώτος όρος που νομίζω ότι το υπενθυμίσαμε και πριν μιλάμε για φορητότητα και όχι πρόσβαση διασυνοριακή. Και αυτό έχει και επιπτώσει. Δηλαδή, στόχο είναι οι χρήστε, οι συνδρομητέ μια υπηρεσία να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία αυτή όταν ταξιδεύουν, όταν ταξιδεύουν σε μια άλλη χώρα τη Ένωση. Όχι όμω ότι ένα ταξιδιώτη που περνά από μια χώρα ε, θα μπορούσε να πάρει μια συνδρομή μια εδαφική υπηρεσία που ε, δεν θα υπήρχε στη δική του χώρα και από τη στιγμή που γυρίζει σπίτι του να έχει πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ τη διασυνοριακή φορτότητα και τη διασυνοριακή πρόσβαση. Η πρώτη κατάσταση θα μπορούσε να ρυθμιστεί με την πρόταση κανονισμού και αυτό το πλάσμα δικαίου, ενώ η δεύτερη ε, κατάσταση ασυνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματική ιδιοκτησία αν δεν υπάρχει αυτή η πολυεδαφική άδεια παροχή υπηρεσιών αλλά δεν είναι τόσο σαφή η διαχωριστική γραμμή στον κανονισμό και πρέπει να διευκρινιστεί η κατάσταση ώστε το κείμενο να μην, οδηγηθεί, ε, να μην ε, βοηθήσει να υπάρχει παράκαμψη της αρχής και να επιτρέπεται τελικά η διασυνορική πρόσβαση ε, σε υπηρεσίες χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Δεύτερη προϋπόθεση, δεύτερος όρος που απορρέει από αυτή την ανάγκη διευκρίνησης της αρχής της φορητότητας σε παραβολή με την πρόσβαση είναι ο προσωρινός χαρακτήρας ε, της διαμονής στο εξωτερικό. Πρόκειται για κεντρικό όρο, κεντρική προϋπόθεση για να γίνει διάκριση ακριβώς μεταξύ πρόσβασης και φορητότητας της συνορικής. Αν δεν υπάρχει όριο σε αυτό το, στην προσωρινή διαμονή και αυτό είναι στη δεκτική ευχέρεια, ε, τότε θα μπορεί να υπάρξουν αποκλίνουσε ερμηνείε και απόψει ό,τι αφορά και τι υπηρεσίε και θα υπάρξουν και καταχρήσει ενδεχομένω. Ξέρω ότι είναι δύσκολη συζήτηση και ήδη υπάρχουν περιχαρακωμένες απόψεις, αλλά για εμάς νομίζω ότι είναι σημαντικό το εύρος, το πεδίο εφαρμογή του κειμένου και ιδίω ο προσωρινό χαρακτήρας να ξεκαθαριστεί και θα πρέπει και όλοι οι εμπλεκόμενοι, εμπλεκόμενοι και ενδιαφερόμενοι φόροι, κοινοβούλιο, ε, συμβουλία, αλλά και οι κάτοχοι δικαιωμάτων, εκπρόσωποι καταναλωτών, πάροχοι περισσότερων να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαβούλευση. Θα πρέπει επίσης να οριστεί καλύτερα το κράτος διαμονής. Κεντρική επίσης έννοια, το είπε και η Μαρία όταν παρουσίασε την πρόταση αυτή και μίλησε για ένα τρίγωνο και ήταν η δεύτερη γωνία του τριγώνου. Αυτό το πλάσμα δικαίου ουσιαστικά το διασυνορικό χαρακτήρα της κατανάλωσης τον διαγράφει και αυτή την ε, κατανάλωση την συνδέει στο κράτος συνήθως διαμονής. Άρα πολύ σημαντικό να οριστεί, πολύ σαφώς αυτός ο όρος. Φαίνεται ότι το Συμβούλιο έχει ήδη σημειώσει πρόοδο τα φορά τον ορισμό αυτό. Προτείνει να γίνεται αναφορά σε ένα κράτο μέλο όπου ο συνδρομητή ε, διαμένει σταθερά ε, και επανέρχεται σε τακτά διαστήματα. Νομίζω ότι είναι λογική, ε, ένα λογικός ορισμός. Αλλά και το κοινοβούλιο νομίζω ότι πρέπει να δραματίσει ένα ρόλο. αφορά Τώρα, ε, το επόμενο που θέλω να πω, τέταρτη προϋπόθεση και απορρέει από τους δύο ορισμούς, ε, κράτος ε, μέλος διαμονή και προσωρινό χαρακτήρα. Να ενισχύσουμε του δύο ορισμού δεν έχει και τόσο νόημα αν δεν υπάρχει δυνατότητα επαλήθευση. Άρα, τέταρτη προπόθεση, επαλήθευση του κράτου μέλου και του προσωρινού χαρακτήρα τη διαμονή. Πρόταση κανονισμού λοιπόν. Ή υποχρεώνει τους παρόχους υπηρεσιών ε, σε αυτή τη φορητότητα, αλλά το κείμενο της Κομισιόν δεν επιβάλλει την επαλήθευση των ε, όρων και προϋποθέσεων. Σε αυτή τη φάση η πρόταση της Κομισιόν λοιπόν χωλαίνει και θα πρέπει να συμπληρωθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το κείμενο λοιπόν πρέπει να προβλέπει υποχρέωση και επαλήθευσης. Και αυτό θα πρέπει να είναι στην τακτική ευχαίρεια των ε, παρόχων υπηρεσιών με μια συμβατική συμφωνία, γιατί ε, δεν υπάρχει και με τους κατόχους των δικαιωμάτων και τις ε, υπηρεσίες ίσως ένας δίκαιος συσχετισμός δυνάμεων το κείμενο ε, είναι άμεσα εφαρμοστέο, δεν, υπάρχει δηλαδή μεταβατική περίοδος, άρα θα πρέπει να προβλέπονται όλες οι παράμετροι υλοποίηση για να μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα ο κανονισμός και μάλιστα κατά τρόπο ομοιόμορφο από όλους τους ε, φόρους. Αυτός είναι και ο στόχος άλλωστε ενός κανονισμού. Παναλαμβάνω λοιπόν επαλήθευση, πραγματική επαλήθευση της διαμονής, του προσωρινού χαρακτήρα, της παρουσίας ενός ε, ταξιδιώτη σε μια άλλη χώρα μέλος. Αυτό θα πρέπει να είναι επίσης μια υποχρέωση για τους παρόχους υπηρεσιών και δεν θα μπορούν να παρεκκλίνουν τι υποχρέωση ε, τη συμβατική οδού. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για την άμεση εφαρμογή αυτή τη ε, αυτού του κανονισμού. Θα πρέπει στον κανονισμό να ορίζονται και τα αποτελεσματικά ε, μέσα της επαλήθευση. Υπάρχει σχετική απόφαση του Συμβουλίου, ίσως σε παράρτημα. Αλλά αυτά τα μέσα θα πρέπει να θεσπίζονται ξεκάθαρα στον κανονισμό και δεν θεωρώ ότι θα ήταν σκόπιμο να εφαρμοστεί εδώ η διαδικασία της επιτροπολογίας γιατί νομίζω ότι είναι μια πολύπλοκη και αδιαφανής ε, διαδικασία για τους ε, φορείς και δεν θα διευκολύνει την άμεση εφαρμογή. Κοινοβούλιο και Συμβούλιο λοιπόν πρέπει να εξετάσουν, να συζητήσουν το κείμενο ε, και να πάρουν όλο τον χρόνο που του χρειάζεται, γιατί στη μελέτη αντικτύπου τη Κομισιόν δυστυχώ δεν θα βρουν τι απαντήσει στι απορίε που μπορεί να γίνουν αυτό το κείμενο. Άκουσα τη Μαρία που εξήγησε ότι ακόμη απομένουν οριστούν αρκετά και λυπούμε που δεν έχει ήδη γίνει αυτό. Γιατί δεν περιλαμβάνονται αυτοί οι στο αρχικό κείμενο. Πριν ολοκληρώσω, ε, θα ήθελα να αναπτύξω μια άλλη σημαντική πτυχή τη παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών προστατευόμενων περιεχομένων, αναθεώρηση τη οδηγία για τι ε, υπηρεσίε οπτικοακουστικών μέσων. Θα κατατεθεί σύντομα από την Κομισιόν η σχετική πρόταση και ελπίζω ότι θα ενισχύσει ε, τις υποχρεώσεις προώθησης των ευρωπαϊκών έργων. Δεν έχω όμως χρόνο για να επεκταθώ πάνω σε αυτό. Ολοκληρώνοντας, υπενθυμίζω ότι ο πολιτικός στόχος αυτής της πρότασης είναι κατανοητός ότι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα μπορούν να καταναλώνουν περισσότερα προστατευόμενα έργα, ταινίες, ε, τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ κτλ. χωρίς ε, περιορισμό λόγω των συνόρων. Ποιο είναι όμως το ζήτημα ότι οι δημιουργοί ε, των τίνων αυτών, ε, των ντοκιμάντερ, δεν θα πληρωθούν παραπάνω. Δεν προβλέπεται κάτι σχετικό. Άρα εμείς θεωρούμε ότι αυτή η νομοθετική πρόταση θα πρέπει να συμπληρωθεί το στομότερο δυνατό με μια άλλη νομοθετική πρόταση που θα αποσκοπεί στην εισαγωγή ενός δικαιώματος αμοιβή για τους δημιουργούς αφόσον είναι τα έργα τους ε, προσβάσιμα σε επιγραμμικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Uh, thank you Ευχαριστούμε. Και τώρα, η κυρία Σαρλότ Λουν Τόμσεν, νομικός σύμβουλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ενώσεων Παραγωγών Ταινιών Κινηματογράφου και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Βίντεο. Δέκα λεφτά, κυρία μου. Ευχαριστώ. Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω στην Ακρόαση και σας ευχαριστώ που την οργανώνετε. Είναι πολύ κατάλληλη φωνική στιγμή οι συζητήσει ε, προχωρούν στην ομάδα εργασία του Συμβουλίου και στο Κοινοβούλιο, σε διάφορε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ οι οποίε εργάζονται για την αναθεώρηση τη ε, πρόταση. Εγώ εκπροσωπώ του ε, παραγωγού ταινιών ε, της Ομοσπονδίας ΦΙΑΠ για όλους τους Ευρωπαίους παραγωγούς και για όλους όσους διανέμουν ταινίες και στο ίντερνετ και σε σε σινεμά. Να σε υπενθυμίσω όλους ότι η ταινία, ο κινηματογράφος είναι η έβδομη τέχνη. Είναι ψυχαγωγία, ε, είναι έκφραση, είναι πολιτισμός. Κάθομαι δίπλα στην εκπρόσωπο της ε, οργάνωσης ε, δημιουργών και πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι ταινίε είναι μια συλλογική δουλειά. Δημιουργούνται γιατί οι διευθυντές, οι δημιουργοί οι ηθοποιοί, τα ταλέντα, το συνεργείο, η παραγωγή, η διανομής, ε, οι διαφημιστές, όλοι αυτοί συνεργάζονται για να φτάσει αυτή η ταινία στο κοινό. Ε, πολλοί άλλοι εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, αλλά κάθε μία από αυτέ τι ομάδε που σας ανέφερα χρειάζεται και χωρίς τη συνεισφορά τους δεν θα υπήρχαν οι ταινίε και οι ταινίε θα φτάνουν ποτέ στο κοινό. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί το σύστημα νεματικών δικαιωμάτων της Ευρώπης ε, εξασφαλίζει αυτή τη δημιουργία ε, και τη δημιουργικότητα και την ε, καλλιτεχνική έκφραση, αλλά και βοηθίζει να εξασφαλίσουμε την ε, επένδυση στην, για την παραγωγή και τη διανομή. Δημιουργεί θέση απασχόλησης και συνεισφέρει στην οικονομία μας. Ο ευρωπαϊκός κλάδος οπτικοακουστικός δίνει 1,2 εκατομμύρια θέσει απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν θέλουμε λοιπόν να εξυγχρονίσουμε το ευρωπαϊκό copyright, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι συνεχίζουμε να επιτρέπουμε την ε, δημιουργία αλλά και την επένδυση. Επίσης, συνεχίζουμε να εξασφαλίζουμε την ε, δυνατότητα ανάκτησης αυτής της, αυτών των ποσών, ας πούμε, ε, της επένδυσης. Η Σεσίλ μίλησε για την πληρωμή φυσικά όλων των, δικαιωμάτων, των κατόχων δικαιωμάτων, που είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Φυσικά δεν κάνουμε ταινίε για πλάκα αλλά για να τα, να τα δει κάποιο, τις ταινίες αυτές για να τις δει κάποιος, κάποιο κοινό. Επομένως, θα πρέπει ε, από την άλλη να υπάρχει το δίκαιο ε, πνευματικών δικαιωμάτων, ούτως ώστε ε, η καλύτερη δυνατή πρόσβαση στο κοινό να εξασφαλιστεί. Ε, μην ξεχνάτε ότι η Ευρώπη ακόμη δεν είναι ένα, μια ανοιχτή ήπειρος και μπορεί η ευρυζωνικότητα να βελτιωθεί, η ταχύτητα της ευρυαζώνης να βελτιωθεί και να έχουμε και καλύτερο νομικό πλαίσιο για το καλό του κοινού, αλλά και των επιχειρήσεων που προσπαθούν να φτάσουν ε, στο κοινό και να καλύψουν τις ανάγκες και τη ζήτηση του κοινού. Είμαι εδώ σήμερα για να σας μιλήσω για την άποψη των ε, διανομέων και παραγωγών ταινιών. Υπάρχει βέβαια το θέμα της φορητότητας από ευρύτερη σκοπιά. Ε, μετά από τα όσα είπε η Σεσίλ, ότι είναι σημαντικό η φορητότητα να παραμείνει φορητότητα και τίποτα παραπάνω. Εγώ θα μιλήσω για πιο, κάτι πιο εστιασμένο. Από την άλλη θα πρέπει να έχουμε την εμπορική ελευθερία για να συλλέγουμε ας πούμε χρηματοδότηση ε, από διάφορες περιοχές, γιατί χρειάζεται αυτό για τη δημιουργία μιας ταινία. Κάθε ταινία έχει το δικό της επιχειρηματικό πλαίσιο, τη δική της οικονομική πραγματικότητα ε, και θέλω να σας δείξω γιατί είναι τόσο σημαντικό να συνεχίζουμε να διατηρούμε την ε, εμπορική και συμβατική ελευθερία για να υπάρξει αυτή η χρηματοδότηση μέσω της ε, διεθνούς συνεργασίας. Χρειαζόμαστε και εσά που παίρνετε αποφάσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ε, αλλά πρέπει, επειδή εδώ διακυβεύονται θέσει απασχόληση, η πολιτιστική και γλωσσική επικοινωνία τη Ευρώπη, εσεί να πάρετε σωστέ αποφάσει. Είναι σημαντικό και για την παραγωγή και για τη διανομή. Ο καθένας έχει τις απόψει του για το αν οι αλλαγέ αυτές θα επηρεάσουν έτσι ή αλλιώς. Το θέμα είναι να είμαστε σίγουροι όμως για να δράσουμε με υπευθυνότητα. Είναι σημαντικό να προχωρήσετε με αποδεικτικά στοιχεία στα χέρια σας και είμαι εδώ για να σας βοηθήσω, ελπίζω, να καταλάβετε λίγο περισσότερο τις λεπτές αλληλεσυνδέσεις ανάμεσα στο, στη χρηματοδότηση, επένδυση δηλαδή και στο, τη δημιουργία. Σας έχω εδώ κάποια παραδείγματα για τον τρόπο που έχουμε συλλέξει χρηματοδότηση, ούτω ώστε να φτιάξουμε κάποιες πρόσφατες ε, ευρωπαϊκές ταινίε. Ε, θα έχετε συνεχεία και την παρουσίασή μου σε χαρτί για να, να δείτε. Η Μαρία αναφέρθηκε στη δική της παρέμβαση στην ε, στο πρόσφατο κείμενο της Κομισιόν, όπου υπάρχει μια αναφορά στην, στο σεβασμό των δικαιωμάτων των δημιουργών στο οπτικοακουστικό τομέα. Επίσης αναφέρθηκε στην πρόταση μιας, της Κομισιόν για βαθμιαία προσέγγιση, ούτως ώστε να υπάρχει πλήρης διεσορυναρική πρόσβαση, που είναι όμως ένας απότατος στόχος. Αυτό κατάλαβα από την ανακοίνωση που εκδόθηκε τον Δεκέμβρη του 2015. Τι σημαίνει να σεβόμαστε τα δικαιώματα των δημιουργών στον κάθε τομέα και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε και αν αυτό παντρεύεται με την πλήρη πρόσβαση. Αυτό θα πρέπει να το δούμε μαζί τους επόμενους μήνες και χρόνια και να αποφασίσουμε γι' αυτό. Αναγνωρίζετε γενικά ότι δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο για να, υπάρχει, να πάρει κανείς άδεια σε διάφορες χώρες. Και το θέμα είναι, δεν είναι αν το θέμα είναι αν είναι οικονομικά σκόπιμο σήμερα. Εμείς ε, στις ταινίε προσπαθούμε για να φτιάξουμε μια ταινία να συγκεντρώσουμε χρηματοδότηση σε διάφορες χώρες. Εδώ έχω αναφέρει κάποια παραδείγματα. Θα ξέρετε διάφορες ταινίε από αυτές. Ίσως δεν έχετε σκεφτεί πριν από τη σημερινή συζήτηση το budget, τον προπολογισμό που χρειάζεται μια ταινία, σαν και αυτές. Ε, είναι από, στις ταινίες που σας έχω βάλει, χρειαζόμαστε από 4 έως 15 εκατομμύρια ευρώ. Επειδή είναι ακριβή μια ταινία για να γίνει, θα πρέπει να υπάρξουν πολλαπλές ε, συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο για να συγκεντρωθεί αυτό το ποσό. Καταρχάς, υπάρχουν συμπαραγωγές. Και όλα τα παραδείγματα, ε, όλες οι ταινίες αυτές είναι ε, συμπαραγωγές συμπαραγωγές Βασιλείου Ελλάδας, Γαλλίας, Γερμανίας, Δανίας, Τσεχίας. Αλλά έχουν και ένα μεγάλο στοιχείο ε, πώλησης, προπόλησης δικαιωμάτων. Βλέπετε εδώ σε εκατομμύρια και βλέπετε και τι ποσοστό του προπολογισμού είναι, που σε αυτήν την περίπτωση είναι ανάμεσα στο 31% ε, και στο 47%. Σε όλες τις περιπτώσεις μιλάμε και πολλά ε, εκατομμύρια ευρώ προπόληση δικαιωμάτων. Και στην τελευταία στήλη ε, θα πρέπει να ανακτήσουμε όχι μόνο τα έξοδα παραγωγής, αλλά και το κόστος του μάρκετινγκ και της διανομής. Επομένως, σε κάθε περίπτωση ε, έχουμε το κόστος της παραγωγής συν έξτρα κόστη. Επομένως, ποιος είναι ο ρόλος των διανομέων σε αυτή την περίπτωση. Θα πρέπει το τελικό προϊόν, την ταινία, να το πάνε, να, την, να το πάρουν και να δημιουργήσουν μια τοπική αγορά σε ξένες χώρες. Παραδείγματο χάρη, ε, έχουμε μια δανέζικη τσεχική συμπαραγωγή στην, ε, βασιλική υπόθεση. Είχε τεράστια επιτυχία στη Γαλλία αυτή, η ταινία. Περίεργο είναι βέβαια, ναι, αλλά είχε. Αλλά ο τοπικό διανομέ διανομέα στη Γαλλία έκανε θαυμάσια δουλειά, προώθησε πάρα πολύ την ταινία και έπεισε το γαλλικό κοινό να πάει να δει αυτή την ταινία, τη βασιλική υπόθεση. Αυτή η δυναμική, αυτή η χρηματοδότηση, οι ανάγκε τη αγορά δεν μπορούν να αλλάξουν μόνο με την επιβολή κάποιων δομών για την αδειοδότηση ή περι, περιορίζοντας την συμβατική ή εμπορική ελευθερία. Και εσείς εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να γνωρίσατε αυτές τις πραγματικότητες στην έκθεση που κάνατε πέρυσι το καλοκαίρι για την εφαρμογή της οδηγίας για τα πνευματικά δικαιώματα. Σας συγχαίρω για αυτό το κείμενο και θα πρέπει να το λάβετε υπόψη. Όταν κοιτάξουμε ειδικά την φορητότητα τώρα, η συνάδελφος ήδη ανέφερε διάφορα από τα προβλήματα και μελήματα που έχουμε ε, και που θα πρέπει μαζί να κοιτάξουμε ούτως ώστε η φορητότητα να παραμείνει φορητότητα. Δεν θα ξαναμπώ σε αυτά τα επιχειρήματα. Θέλω να προσθέσω όμως ότι όλα τα στοιχεία υπάρχουν εδώ, τα έχετε στη διάθεσή σας και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η πρόταση ε, συνάδει με το διεθνές δίκαιο και την υποχρέωση που, ή τις υποχρεώσεις που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση διεθνώς. Τώρα, για το πώς θα προχωρήσουμε για να μην ξεχνάμε και το χρόνο. Η σημασία τη εμπορική ελευθερία είναι τεράστια για να συγκεντρωθεί η χρηματοδότηση, για να γίνει το καλύτερο μάρκετινγκ, Ε, Επίση, θα πρέπει οι νομικέ υπηρεσίε να είναι κατάλληλε. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να δουλεύουμε για να ενημερώνουμε το κοινό μα για το πού μπορούν να βρουν ε, επίση ε, νόμιμο περιεχόμενο. Ε, έχουμε τεράστια επιλογή που καλύπτει τα γούστα όλων. Επίσης, συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες. Εκεί που δεν μπορούμε να κάνουμε κλασική εμπορική διανομή, να δώσουμε εναλλακτικέ λύσεις για να υπάρξει πρόσβαση του κοινού στις δημιουργίε. Και επίσης θα πρέπει να έχουμε μία προσέγγιση πολύ ε, υπεύθυνη, ε, που να βασίζεται σε στοιχεία, ούτω ώστε να διατηρήσουμε τον κλάδο για το μέλλον τη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Thank you, ε, πολύ. Μάγνους Μπρουκ. Διοικητικό Συμβούλιο της ε, Ένωσης Τηλεοπτικών Σταθμών Ευρώπης και έχετε το λόγο. Uh, Θα ήθελα να ευχαριστώ την Επιτροπή σας ε, για την πρόσκληση να μιλήσω εδώ. Είμαι επικεφαλής λοιπόν του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης των Τηλεοπτικών Σταθμών αλλά και της ε, της ρυθμιστικής ε, ε, υπηρεσίας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς παραγωγούς τηλεοπτικού περιεχομένου στην Ευρώπη. Μία από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε από αυτή την πρόταση σε σχέση με το ελεύθερο περιεχόμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την ITV λοιπόν η ιδέα ότι ο, Βρετανός πρέπει να έχει, ο Ευρωπαίος πολίτης πρέπει να έχει τη δυνατότητα της πρόσβασης στο περιεχόμενο που έχει πληρώσει όταν ταξιδεύει σε ένα άλλο κράτος έχει βεβαίως να κάνει με τον πυρήνα της ψηφιακής αγοράς και υποστηρίζουμε τη φιλοδοξία. Η ITV εξασφαλίζει και την ελεύθερη online υπηρεσία και την ε, συνδρομητική υπηρεσία στους ε, πελάτες της. Η τελική μορφή του κανονισμού λοιπόν πρέπει να εξασφαλίζει για τον πάροχο, τον καταναλωτή και τον δικαιούχο ασφάλεια δικαίου. Είναι δύσκολο να αρνηθεί κανεί ότι ο κανονισμό ε, ενώ θα επιτρέπει βεβαίω καταπληκτικό κατα, τεράστιες προκλήσεις συντονισμού θα προσφέρει υπηρεσία στον καταναλωτή μεγάλη αλλά δεν πρέπει να δώσουμε βραχυπρόθεσμα ωφέλη σε ορισμένους χωρίς να καλύψουμε άλλους καταναλωτέ, οι οποίοι ενδεχομένω δεν ταξιδεύουν και έτσι θα βρεθούν σε χειρότερη θέση γιατί αυτό δεν πρέπει να καταστεί αυτός σκοπός. Οι υπηρεσίες λοιπόν που πρέπει να καλύπτονται από τον κανονισμό πρέπει να προσδοριστούν και το δικαίωμα επαλήθευσης. Ο στόχος της πρότασης είναι όταν κάποιος έχει πληρώσει για μια διαγραμμική υπηρεσία να έχει την πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία και όταν ταξιδεύει εκτός της χώρας στην οποία έχει τη συνδρομή. Αυτές οι υπηρεσίες λοιπόν θα πρέπει να καλύπτονται από τον νέο κανονισμό. Η Hub Plus λοιπόν, η υπηρεσία που έχει η ITV, δωρεάν, με 3,99 3,99 λίρες τον μήνα είναι διαθέσιμη στον πελάτη της ITV όταν ταξιδεύει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτείνεται επίσης μη ε, πληρωνόμενα, δωρεάν δηλαδή, δωρεάν περιεχόμενο ή υπηρεσία να προσφέρεται υποχρεωτικά και με, με φορητότητα. Και αυτό σημαίνει ότι ο ορισμός της επαλήθευσης θα ορίσει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Κάποια ασάφεια όμως ως προς τον προσδιορισμό και την, της μπορεί να οδηγήσει σε δωρεάν οπτικοακουστικές υπηρεσίες κατά τρόπο που να αποβαίνει εις βάρος των συμφερόντων όλων των χρηστών αυτών των υπηρεσιών ανεξαρτήτως του ε, που ταξιδεύουν και θα εξηγηθώ. Έχει ένα online catch-up ως σύστημα η ITV, δηλαδή μπορεί να δει κανεί παλαιότερο περιεχόμενο εάν έχει χάσει ένα επεισόδιο και ολόκληρη σειρά ακόμη του Downton Abbey της σειράς αυτής ε, μπορεί να το δει εκ των υστέρων. Είναι βέβαια πολύ δημοφιλής υπηρεσία με 15 εκατομμύρια αιτήματα για ε, να δει ε, περασμένο επεισόδιο ο θεατής μας ένα συγκεκριμένο επεισόδιο του Downtown Abbey. Ε, έτσι λοιπόν κερδίζει σε σχέση με την αγορά ενός ε, σετ DVD ε, ο καταναλωτής και βέβαια πέραν από, το, από κάποιες ε, διαφημίσεις είναι δωρεάν αυτή η υπηρεσία. Ε, δωρεάν περιεχόμενο λοιπόν, ωστόσο ο παρέχον το δωρεάν αυτό περιεχόμενο πιστεύει ότι θα πρέπει ο, ο καταναλωτής που θα έχει αυτή τη δωρεάν υπηρεσία να είναι όσο δυνατόν πιο κοντά στον πάροχο. Αντίθετα με τις, ε, κατά, με τις επιπληρωμή υπηρεσίες δεν συλλέγουμε στοιχεία πιστωτική ιδρύματος ή κάρτας πιστοτικής ε, γιατί μπορεί να αποφύγει ο καταναλωτής να έρθει σε εμάς. Κάποια δεδομένα μόνο ε, για την πρώτη φορά που μπαίνει κανείς σε μια υπηρεσία, μερικές φορές και με σύμβαση με το χρήστη, ώστε η ε, η υπηρεσία να προσφέρεται κατά τρόπο να αποδεκτό και βέβαια να μην υπάρχουν καταχρήσεις. Όνομα, επώνυμο και ε, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δηλαδή καλούμε τα οι καταναλωτέ να δίνουν. Δεν προσπαθούμε βέβαια να επαληθεύουμε τις ταυτότητες κτλ. Αλλά αυτό δεν είναι πάντοτε δυνατόν. Εν γέννη έχουμε κάποια ιδέα του, καταναλω... του ποιος είναι ο χρήστη μας, αλλά δεν είναι απόλυτα σαφής η εικόνα και πάντως δεν έχουμε στοιχεία τραπεζικά και πιστοτικής κάρτας. Γιατί λοιπόν αυτά τα βασικά στοιχεία, γιατί συλλέγονται. Δύο λόγοι. Καταρχάς για να δίνουμε ε, κατά βάση την υπηρεσία που τους φαίνεται, φαίνεται πιο ενδιαφέρουσα, είτε πρόκειται για το ποδόσφαιρο στη Σκοτία ή ένα, ε, μια υπηρεσία ειδησιογραφική. Δεύτερον, για να μπορούμε να κατευθύνουμε διαφημίσεις αναλόγως του ενδιαφέροντος και της καταλληλότητας του καταναλωτή, καλύτερα υπηρεσία, καλύτερη υπηρεσία εν γέννη δηλαδή. Ανησυχία μας είναι ότι σε ορισμένες πιθανές εκδοχές του κανονισμού οι ελεύθερες αυτές υπηρεσίες μπορεί να θεωρηθούν ότι επαληθεύουν την συνήθη κατοικία του χρήστη. Γιατί είναι αυτό το πρόβλημα. Μα γιατί απλώς όταν δεν επιβεβαιώνουμε επαρκώς το, την κατοικία του χρήστη. Δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι λοιπόν με όλη την προσπάθεια και να κάνουμε. Φερρυπίν είχαμε 6.000 χρήστες που ισχυρίζονταν ότι ζουν στο Buckingham, στο παλάτι του Buckingham. 13.000 χρήστες που έδιναν ηλικία άνω των 110 ετών. Αυτά είναι παραδείγματα βεβαίως ακραία ως προς την ταυτότητα των χρηστών, αλλά δείχνουν ότι για να τα επαληθεύσουμε θα χρειαστεί και χρόνο και χρήμα. Πολύ πιο περίπλοκο επίσης θα είναι το να έχουμε ε, δεδομένα ε, βασικά ε, παρόμοια, όπως πολύ με το όνομα John Smith και ηλικία 25 ετών. Θα είναι πολύ δύσκολο να γίνει η επαλήθευση. η κάλυψη μπορεί να αφορά μέχρι και 700 νοικοκυριά. Για να μπορέσουμε λοιπόν να έχουμε την υψηλότερη αξία και το πιο δημοφιλές περιεχόμενο με το Downton Abbey και τη δυνατότητα να δει κανείς περασμένα επεισόδιο το Catch Up Service, αυτό μπορούμε να το προσφέρουμε μόνο στον κάτοικο του Ηνωμένου Βασιλείου. Εάν ανοίξουμε την υπηρεσία αυτή υπάρχει κίνδυνος να μην ε, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ε, εισόδημα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει πολύ μεγάλη αξία εμπορική και άρα θα χάσουμε εισόδημα το οποίο θα ήταν χρήσιμο για περαιτέρω επενδύσεις και νέα, ε, νέο περιεχόμενο. Η πρόσβαση λοιπόν σε ελεύθερες υπηρεσίες δεν θα εξασφάλιζε για όλους τους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι χρήστες μας την ίδια ποιότητα και ταυτόχρονα αυτή η υψηλή ποιότητα θα μπορούσε να χαθεί ακόμη και από την δωρεάν υπηρεσία, από το free to air service μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο, εις βάρος εκείνων οι οποίοι δεν ταξιδεύουν έξω από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και έτσι τότε θα έπρεπε ο καθένας να πληρώνει για να έχει αυτό το βασικό περιεχόμενο στο Ηνωμένο Βασίλειο που ήταν μέχρι τώρα δωρεάν. Δεν νομίζω ότι αυτό θα το δεχθούν οι καταναλωτές. Ε, η φορητότητα λοιπόν για τις επιπληρωμή υπηρεσίες και υψηλή ποιότητα για δωρεάν υπηρεσίες, πώς θα εξασφαλιστεί. Νομίζουμε ότι η μέγιστη ασφάλεια δικαίου θα, ήταν να, θα εξασφαλιζόταν εάν οριζόταν συγκεκριμένα στον κανονισμό ότι οι δωρεάν υπηρεσίες το free to air δεν είναι αυτόματα φορητέ, αλλά ότι μπορεί αργότερα να μπουν με τρόπο εθελοντικό μέσα στον κανονισμό, με ένα σύστημα ε, κούσιας συμπερίληψης. Οπότε, ναι, αλλά μόνο όταν ο ε, πάροχος μπορεί να εξασφαλίσει δυνατότητες συγκρίσιμες για ε, τις ε, συνθήκες που χρειάζεται. Κάθε ε, επαλήθευση λοιπόν θα πρέπει να είναι σωστή και τόσο για τον καταναλωτή, για τον πάροχο και για το δικαιούχο στο, για το πιο δημοφιλές περιεχόμενο που έχει στη διάθεση του δωρεάν το ακροατήριο σε όλη την Ευρώπη. Θα ήταν κρίμα η συνεχιζόμενη ελκυστικότητα και βιωσιμότητα της ε, δωρεάν ελεύθερης ε, τηλεόρασης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να κινδυνεύσει. Έχουμε να κάνουμε τεράστια ε, έκταση και επέκταση επιλογών εκατομμύριων των καταναλωτών στα τελευταία χρόνια που κινδυνεύει βεβαίως. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ. Έχουμε 15 λεπτά για ερωτήσεις ε, μετά από όλες αυτές τις παρουσιάσει που ακούσαμε. Να δώσω καταρχάς το λόγο στους εισηγητές, δηλαδή τον Σαμαρί Καβάντα και τον Μάρκο Ζούλο. Από την Ίμκο και τη Σαμπίνη Φερχάγεν από την Κάλτ. Και μετά βλέπουμε αν μείνει χρόνος και πόσο, Ο Ζάμαρη Καβαντά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω του ε, ομιλητέ. Την κυρία Μαρία Μάρτιν Πρέτσπορτ απ' όλα Πρέπει να πω ότι η συνετή προσέγγιση της Κομισιόν είναι ισορροπημένη. Έχουμε συγκρατημένα αισιόδοξο συνήθως ό,τι αφορά ε, θεσμούς που πρέπει να ελέγξουμε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμίσουμε στην προκειμένη περίπτωση ότι έχουμε και επαγγελματισμό και ισορροπία και όλα αυτά προνίζουν καλά για, το, ε, για την πρόταση αυτή. Λοιπόν, να σας δώσω το δικό μας σκεπτικό. Η διασυνορική φορητότητα ε, αποτελεί ένα ακόμη βήμα για την καταπολέμηση της πειρατείας και αυτό είναι θετικό. Οι Ευρωπαίοι πολίτες που μετακινούνται, που ταξιδεύουν θα μπορούν να συνεχίσουν ε, υπό συνθήκε νομιμότητα να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο το οποίο έχουν αποκτήσει προηγουμένως στη χώρα διαμονή του. Δεύτερον, ο κανονισμό περιφορητότητας θα πρέπει να είναι αναλογικός ε, να προσαρμόζεται δηλαδή στις πραγματικότητες ε, της αγοράς υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και στις πραγματικές ε, ανάγκες των καταναλωτών. Ο αριθμό τώρα των δυνητικών καταναλωτών που θα μπορούν να, μεταφέρουν τις υπηρεσίες τους με βάση τις ενδείξεις θα ήταν γύρω στα 29 άντε 30 εκατομμύρια, 5,7% δηλαδή των Ευρωπαίων καταναλωτών. Άρα είναι ένα θύλακα, είναι μια αποκλειστική μικρή αγορά, είναι μικροαγορές αν θέλετε, που δεν νομίζω ότι θα ταράξουν το βασικό κανόνα, που φυσικά ε, μου είναι ιδιαίτερο προσφυλη. τώρα, ένα άλλο θέμα. Σε ό,τι αφορά διαφορά μεταξύ πρόσβαση και φορητότητας. πάντα για υπηρεσίε υπογραμμικού περιεχομένου. Καταρχά δεν υπάρχει καμία αντίφαση, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, μεταξύ εδαφικότητα και φορητότητα περιεχομένου. Έψαξα, ξανάψαξα και δεν βρήκα. Πού είναι η δυσκολία, τουλάχιστον να κάποιο θέλει να είναι Θεωρώ απλά ότι με τη φορητότητα ο καταναλωτή όταν μετακινείται μπορεί να συμβουλεύεται ένα περιεχόμενο που εκ των προτέρων έχει αποκτήσει, επαναλαμβάνω, σε ένα ε, κράτος, το κράτος κατοικίας του με νόμιμο τρόπο. Νομίζω είναι το στοιχειώδες αυτό. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό. Τώρα, ο καταναλωτής ε, έχει αποκτήσει νομίμως, είπαμε, ε, μια υπηρεσία επικοινωνικού περιεχομένου στη χώρα συνήθω διαμονή του. Και θα μπορεί να συμβουλεύει το περιεχόμενο αυτό όταν μετακινείται προσωρινά στο εξωτερικό. Η απαραίτητη προϋπόθεση αυτής της πραγματικής είναι να μην παραβιάζουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησία. Δηλαδή δημιουργεί να αμείβονται. Γνωρίζουμε ε, πόσο ευάλωτε είναι τα δικαιώματα των ε, δημιουργών και σίγουρα πρέπει να φροντίσουμε να γίνονται σεβαστά τώρα. Η, ε, ο δωρεάν χαρακτήρας, ε, η φορητότητα είναι δωρεάν υπηρεσία. Γιατί είναι νομίζω αναπόσπαστο τμήμα της συνδρομής. Ουσιαστικά πρόκειται για μια τεχνική υπηρεσία που επεκτείνει αυτό το δικαίωμα, το κεκτημένο δικαίωμα, σε μια άλλη χώρα προσωρινά. Οι δικαιούχοι τώρα μπορούν να ε, επαναδιαπραγματευτούν προς τα άνω το συμβόλαιό τους με τους παρόχους υπηρεσιών αν τεθεί σε ισχύ αυτός ο κανονισμός. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Είναι μια βάση. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα το χρονικό όριο, η φορητότητα θα πρέπει να είναι μια παρεχόμενη υπηρεσία, χωρίς κατά την απόψή μου ε, περιορισμό στο χρόνο. Γιατί το αντίθετο θα οδηγούσε σε πειρατεία και σε ασάφεια δικαίου. Επομένως, από τη στιγμή που το κριτήριο περί, ασφαλούς, ε, περί διαμονής ελέγχεται, επαληθεύεται με σοβαρότητα και αυτό πρέπει να προβλεφθεί, δεν ότι χρειάζεται και ότι υπάρχει ανάγκη να μπει ένα χρονικό όριο για τον κατανάλωτη, γιατί η προσπάθεια που θα πρέπει να καταβληθεί πέραν αυτού του ορίου, αν δηλαδή παραταθεί η προσωρινή διαμονή, θα είναι πάρα πολύ δάπανη. Και δεν ξέρω και κατά πόσο μπορεί να ελεγχθεί η ρίστα παρόδο. Τώρα, τα κριτήρια επαλήθευση τη συνήθω διαμονή θα πρέπει να είναι στεναρά, αλλά χωρίς ε, να υπάρχει παραβίαση της ιδιωτικότητας του καταναλωτή από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει αυτή η φορητότητα. Τα δικαιώματα δημιουργού όμω πρέπει, όπω είπαμε, να είναι κεκτημένα. Το πάμε και το ξανάπαμε. Και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να φροντίσουμε φορητότητα να μην διαταράξει την αναδιανομή τη δημιουργική αξία σε βάρο των καλλιτεχνών, δικαιούχων, αλυσίδας παραγωγή. Ε, αυτά σε αντρέ γραμμέ. Μπορούμε να είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε συζήτηση. Παναλαμβάνω όμω ότι είναι αρκετά άρτια και ισορροπημένη η πρόταση τη Κομισιόν να μην έχουμε δράματα ούτε από την πλευρά των καταναλωτών, ούτε από την πλευρά των δικαιούχων και των αλυσίδων παραγωγή. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε. Μάρκο Τζούλο, από την Επιτροπή ΜΚΟ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ του ε, ομιλητέ του πάνελ. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσει προ αυτού. μια και είναι εδώ παρόντε. Αν κατάλαβα καλά, το να προβλέψουμε την φορητότητα του online περιεχομένου για τους καταναλωτές σημαίνει αλλαγή των ε, συμβολέων ανάμεσα στους ε, κατόχους δικαίου, στους παρόχους και στους ε, απλούς καταναλωτές. Πώς θα επηρεάσει αυτό το κόστος των αδειών στο εσωτερικό του κλάδου. Τι κόστος θα συνεπιφέρει αυτό για τους καταναλωτές μια και θα αλλάξουν οι συμβάσει. Θα μειωθεί η προσφορά για τον τελικό χρήστη ή θα αυξηθεί η τελική προσφορά. Νομίζω ότι αυτό το θέμα ε, έχει προκύψει σε πολλές επαφές που έχω κάνει με ειδικού. Το δεύτερο είναι το δωρεάν περιεχόμενο. Όπως υπόθηκε, μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα, οι δωρεάν υπηρεσίες δεν υποχρεούνται να εξασφαλίσουν φορητότητα. Όμως συχνά ο χρήστης πληρώνει την υπηρεσία όχι με λεφτά, αλλά δίνοντας τα δικά του προσωπικά στοιχεία. Είμαστε σίγουροι ότι έχουμε ορίσει σωστά σε αυτήν την περίπτωση τη δωρεάν υπηρεσία, την προσφορά δωρεάν περιεχομένου, εν Κύριε Φερχάινεν, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέροντα όσα ακούσαμε και μάθαμε σήμερα. Η Επιτροπή Πολιτισμού έχει ήδη καταθέσει γνωμοδότηση που είναι σε διαδικασία ε, επεξεργασία. Ε, σημαντικό από αυτά που υπόθηκαν ήταν νομίζω το ζήτημα του κράτους της συνήθους διαμονής, δηλαδή να υπάρχει ένα σαφής ορισμός της, της ε, συνήθους διαμονής και εδώ χρειάζεται ίσως πιο αυστηρή διατύπωση, πιο συγκεκριμένη διατύπωση. Και νομίζω ότι, όπω το έχω προτείνει και μέσα στη γνωμοδότηση, μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη συνέχεια και με μια διαδικασία με κατεξουδότηση πράξη να ε, επαληθεύει αν όντω το νομικό πλάσμα αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε ισχύει αν τυχόν είναι κενό περιεχομένου. Υπάρχει λοιπόν αυτό το πλάσμα δικαίου ότι έχει κανείς στο κράτος ε, της ε, ηθαγένειας ε, αποκτήσει το δικαίωμα σε πρόσβαση σε ένα περιεχόμενο και βέβαια το θέμα είναι αν μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό το δικαίωμα και πέραν αυτού του, του κράτους και έξω από το κράτο, Αλλά βέβαια το ζήτημα είναι με το, νομικό, με το πλάσμα δικαίου αυτό να μην γίνεται αλλίωση τη σύμβαση, να μην εισαχθεί δηλαδή ένα νέο μοντέλο επιχειρησιακό ε, ή συμβατικό, αλλά να υπάρχει δυνατότητα τα δικαιώματα αυτά να τα χρησιμοποιεί κανεί και σε μια άλλη χώρα Υπηρεσίε και άλλε μάλιστα, όχι μόνο τηλεοπτικό περιεχόμενο αλλά και βιβλία κτλ. Αυτό ακριβώ. και νομίζω η τεχνική προσαρμογή, αυτό που λέγαμε με την ε, μεταβατική περίοδο, θα έχει να κάνει με την επαλήθευση των συμβάσεων. Και για να αναφερθώ και στο όσα είπε ο συνάδελφος πριν, ε, η δωρεάν τηλεόραση, το free to air, έτσι, όχι η δημόσια, δεν έχει να κάνει με σύμβαση με τον χρήστη και άρα δεν υπάρχει περίπτωση επαλήθευσης της κατοικίας του χρήστη, των δεδομένων του χρήστη προκειμένου να υπάρξει αυτή η φορητότητα και άρα δεν υπάρχει υποχρέωση για παροχή της υπηρεσίας. Εάν όμως κάνετε επαλήθευση τότε θα πρέπει με βάση τη διοσύνη του κανονισμού να προσφέρετε και την φορητότητα. Επομένως, η ε, επαλήθευση και η ταυτοποίηση του ατόμου του χρήστη συνδέεται άμεσα με τη φορητότητα. Πράγμα το οποίο για μένα δημιουργεί κανένα πρόβλημα, απλώς και μόνο άπαξ και γίνει η επαλήθευση της ε, χώρας ε, της συνήθως διαμονής. Έχουμε και την φορητότητα. Ε, βέβαια, η επαλήθευση δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε διαρκώς με ένα σύστημα tracking των ε, χρήστη, να βλέπουμε που βρίσκεται, τι βλέπει και όλα αυτά. Έτσι λοιπόν ε, θα πρέπει να παραμείνει, και αυτό το απευθύνω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, να παραμείνει ανοιχτό το ζήτημα. Δηλαδή να εξετάσετε το αν κάποιο απλώς δεν είναι στην ε, συνήθη διαμονή του. Θα πάρω για παράδειγμα τον οδηγό του φορτηγού, ο οποίος σε κάποιο κράτος μέλος έχει συνήθη διαμονή, αλλά ταξιδεύει πάρα πολύ. Δεν με νοιάζει να δω πόσες μέρες το μήνα ή τη βδομάδα λείπει από το σπίτι του, αλλά θέλω να μπορεί όταν είναι μέσα στην, στο κουβούκλιο του φορτηγού του να παρακολουθεί το περιεχόμενο για το οποίο έχει συνάψει τη σύμβαση. Δεν θέλουμε φυσικά να γίνεται αυτό το tracking, η παρακολούθηση της παρουσίας ημί του ε, καταναλωτή. Πρέπει να, γίνει, να εξασφαλιστεί απόλυτη προστασία των προσωπικών δεδομένων και πιστεύω ότι με την πρόσθεση της Επιτροπής θα το καταφέρουμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και τώρα Έχουμε ελάχιστο ελάχιστο χρόνο και παρακαλώ όποιον από τους προσκεκλημένους έχει πρόθεση να απαντήσει σε ερωτήσεις που του έχουν απευθυνθεί να λάβει το λόγο. Μας μένει ένα λεπτό ουσιαστικά. Thank you um, um, Ευχαριστώ πολύ. Στο ζήτημα του κυρίου Σούλα, της κυρίας Φερχάιεν, για το επαμοιβή ή δωρεάν περιεχόμενο. Είπα και στην ε, εισαγωγή μου, θα το επιβαλθεύσει φαντάζομαι και η Μαρία, ότι δεν υπάγονται όλες οι υπηρεσίες, το free-to-air παραδείγματι ή δωρεάν, το δωρεάν περιεχόμενο δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Αλλά βέβαια άλλη συζήτηση είναι το να υπάρχει μια σύμβαση όπου προσφέρεται κάτι άλλο ως αντάλλαγμα. Και ίσως αυτό θα πρέπει να το εξετάσουμε μαζί με όλη τη στρατηγική της Επιτροπής και την άλλη πρόταση που επίσης έχει να κάνει ε, η οποία επίσης το Δεκέμβριο για το ψηφιακό περιεχόμενο που τώρα αρχίζουν να αναπτύσσονται δικαιώματα για καταναλωτές σε συμβάσεις όπου ο καταναλωτής δίνει ένα άλλο αντάλλαγμα, όχι όπως υπερδείγματι προσωπικά δεδομένα. Άρα, όταν προσφέρω για να έχω πρόσβαση σε δεδομένο, σε περιεχόμενο, πρόσβαση σε προσωπικά μου δεδομένα ή άλλο ε, στοιχείο μου, τότε μήπως θα έπρεπε να έχω και εκεί το δικαίωμα της, προσβατώ, της ε, φορητότητας. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. Για μένα είναι σαφές όταν υπάρχει μια σύμβαση για κάποιες υπηρεσίες τότε πρέπει να καλύπτονται. Εάν καλύπτονται, εάν κάποιος θέλει να καλύπτονται τότε θα πρέπει να τις ε, καθιστά, ε, να εξασφαλίσει τη δωρεάν προσβασιμότητα κτλ. Η κυρία Πράτ νομίζω ήθελε το λόγο. Ναι, Πρόεδρε, και στο συγκεκριμένο αυτό σημείο. Όπως πει η κυρία Φερχάιεν, όντως, δωρεάν υπηρεσία δεν υπάρχει. διάκριση στον κανονισμό γίνεται όχι μεταξύ δωρεάν και μη δωρεών, δωρεάν ή ε, μη υπηρεσιών, αλλά υπηρεσιών που, που προσφέρονται έναντι ε, χρηματικού ανταλλάγματος ή άλλου τύπου. Όπως, για η διαφήμιση αντάλλαγμα. Στη διαφήμιση προσφέρεται ο χρόνος του καταναλωτή. Έτσι λοιπόν γίνεται διάκριση με βάση αυτά στον κανονισμό και οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται με αντάλλαγμα χρηματικό αυτόματα μπαίνουν στην φορητότητα με επαλήθευση της συνήθους διαμονής. Αντίθετη είναι η κατάσταση στις υπηρεσίες ε, για τις οποίες ε, δεν απαιτείται αντάλλαγμα χρηματικό όπου μπορεί να γίνει η επιλογή της συμπερίληψης σε αυτές τις υπηρεσίες, το opt το λεγόμενο και αυτό, γιατί για μας υπάρχει ζήτημα αναλογικότητας και τελικού συμφέροντας συμφέροντος του καταναλωτή. Ακούσατε σε τελευταία ανάλυση την επιχειρηματολογία της ITV, ότι δηλαδή κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες δεν υπησέρχονται σε επαλήθευση της διαμονής του καταναλωτή. Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για υπηρεσίες του οπτικοακουστικού τομέα που άλλωστε δεν προσφέρουν καν περιορισμό για το περιεχόμενο όπου βρίσκεται κανείς αναλόγως του που βρίσκεται κανείς και κατά πάσα πιθανότητα η αυτόματη επαλήθευση που θα επέβαλε ο κανονισμός σε μια τέτοια περίπτωση για το free-to-air θα ήταν είτε εις βάρος του καταναλωτή είτε εις βάρος ενός μηχανισμού επαλήθευσης για τους λοιπούς χρήστες που είναι ο βασικός στόχος του κανονισμού και πάλι δεν αποκλείονται τα περιεχόμενα και χρήσεις αυτή, ε, μπορούν να συμπεριληφθούν αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Και εσείς. Και βεβαίω υποστηρίζουμε σε αυτό την ε, θέση της Επιτροπής. Το κρίσιμο είναι η επαλήθευση. όχι αν ε, πρόκειται για πολλά ή λίγα δεδομένα, όταν υπάρχει σε νομικούς, με την νομική έννοια του όρου σύμβαση σημαντικό εν είναι η υπηρεσία που προσφέρεται και δεν μπορεί να επαληθευτεί για το free-to-air ε, το ε, θέμα της σύνδεσης διαμονής ή τα λοιπά στοιχεία. Ε, εν γέννη, οι λοιποί πάροχοι έχουν σύμβαση με τον χρήστη και πολύ καλά κάνουν. Ωστόσο και σε διαδραστικές υπηρεσίες υπάρχουν όροι χρήσεως που επιβάλλονται κατά τρόπο συμβατικό με τη χρήση δηλαδή της υπηρεσίας αποδέχεται κανείς και τους όρους της σύμβασης και είναι δωρεάν. Ε, νομίζω ωστόσο ότι γίνεται η βασική διάκριση όπως και από την Επιτροπή δηλαδή της καταβολής χρηματικού αντιτιμού και ε, άρα υποβολή στοιχείων πιστοτικής ε, τράπεζας ε, ή τραπεζικού λογαριασμού και εκείνων που δεν απαιτούν. Βέβαια ένας καταναλωτής ο οποίος πηγαίνει σε μια δωρεάν υπηρεσία δεν θα θέλει να δώσει τα στοιχεία της επιστατικής του τρα... Ε, κάρτας ή του τραπεζικού λογαριασμού που μετά θα μπορούσαν να μετατρέψουν την υπηρεσία σε επί αμοιβή. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Δυστυχώ έχει εξαντληθεί ο χρόνο μα. Ευχαριστούμε του διερμηνεί για την υπομονή του. Ο κύριο Καβαντά θα κάνει μια πολύ στομή δήλωση μόνο. Ευχαριστώ, πρόεδρε, και δεν θέλω να καθυστερήσω το συναδέλφους και το μεσημεριανό τους πρέπει νομίζω να μας απασχολήσει στο πρόσθετο αυτό περιεχόμενο που προσφέρεται και το μέλλον των ε, παραδοσιακών δημοσίων υπηρεσιών οπτικού ακουστικού υλικού στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι καθόλου δεδομένο και θέλω να πω προς τους συναδέλφους αλλά και όλους τους ομιλητές ότι και η ομάδα μου και εγώ είμαστε στη θέση σας και θα παρακολουθήσουμε πολύ μεγάλη προσοχή κάθε ζήτημα που θα μπορούσε να ενδιαφέρει ε, στην υπόθεση αυτή γιατί θέλουμε να κάνουμε στο δυνατόν καλύτερη δουλειά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Πρόεδρος ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη από τους αδέλφους που θέλησαν να λάβουν το λόγο αλλά δεν μπόρεσαν. Ασφαλώς θα δοθούν και άλλες ευκαιρίες για να επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ τους προσκεκλημένους μας και τους διερμηνείς λίγο, Πρόεδρος για τον επιπλέον χρόνο που μας προσέφεραν.